Goedemorgen ehm, Καλή μέρα κυρίες και κύριοι. Ο Γιάνν Βίλτ δεν είναι εδώ σήμερα, ζητά συγγνώμη, δεν ε, μπορούσε δυστυχώς να είναι παρόν. Οπότε αναλαμβάνω εγώ να τον αντικαταστήσω όσο καλύτερα μπορώ. Έχουμε μια πυκνή μερίσια διάταξη, έχουμε και από την Επιτροπή, καλώς ήρθατε, Έχουμε κάποιες ερωτήσεις για σας κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που είσαστε εδώ. Πρώτα απ' όλα όμως πρέπει να ψηφίσουμε, ζητούμε συγγνώμη για αυτό, είναι μια μικρή ψηφοφορία που έχουμε να κάνουμε. Και μετά μπορείτε να έρθετε εδώ πιο κοντά, να μας μεταφέρετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Συμφωνείτε όλοι? Συμφωνείτε όλοι με την ημερήσια διάταξη, με το σχέδιο. Δεν έχετε καμιά αλλαγή να ζητήσετε, τίποτα ωραία. Στη συνέχεια, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Καλά τις γλώσσες, ότι είμαστε web streamed. Ψηφίζουμε μετά ηλεκτρονικά. Ελπίζω να έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες σας, γιατί μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη η ψηφοφορία. Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό ως ανακοινώσει του Πρόεδρου είναι όλη η συζήτηση που κάνουμε εδώ και μήνες και χρόνια με το Συμβούλιο για την απαλλαγή. Νομίζω ότι είναι γνωστό το θέμα, είναι γνωστό που υπάρχουν διαφωνίες. Κάποια στιγμή είχαμε στείλει και μια επιστολή στον Επίτροπο Σεμέτα, ζητώντας του ενημέρωση για την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 25 Νοεμβρίου ήταν η επιστολή αυτή. Στην συνεδρίαση των ε, συντονιστών στις 29 Νοεμβρίου εξετάσαμε την ε, απάντηση και οι συντονιστές εξέφρασαν την επιθυμία ο Επίτροπος Μέτα να έρθει και να μας ενημερώσει. Οπότε κύριε Επίτροπε, στο σημείο 4 να ξεκινήσετε εσείς για να μας παρουσιάσετε τη θέση της Επιτροπής όσον αφορά την απαλλαγή του Συμβουλίου. Να μας ενημερώσετε σχετικά με αυτή την επιστολή της 25ης Νοεμβρίου. Σύμφωνοι? Καλώς. Οπότε ξεκινάμε την ψηφοφορία. Πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Έρενχάουσερ. Είναι η πρώτη του, ε, συγχαρητήρια. Πρόκειται για τον δημοσιονομικό έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας που διαχειρίζεται η ΕΚΟ. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Δεν ξέρω ο κύριος Έρνχάουζεν που θέλει να πει κάτι προηγουμένως. Όχι. Ωραία. Οπότε αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Έχετε τον κατάλογο μπροστά σας, ελπίζω. ψηφίζουμε πρώτα το σημείο 4, τροπολογία αριθμό 1 του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 2. Βάιλερ και Μπέρμαν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 3. Βάιλερ Μπέρμαν. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4, Ερενχάουζερ, είναι συμβατή με την τροπολογία 3 ως προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ. Κα... κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 5, Ehrenhauser υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 παράγραφος, τροπολογία 6, Ερνχάουζερ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 7, Μπέρμαν και Βάιλερ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρα στις ψηφοφορίες. Αποτέλεσμα. 7 υπέρ, 4 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Παράγραφος 9, τροπολογία 8. Χάρτογκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 10, τροπολογία 9. Βάιλερ Μπέρμαν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11, τροπολογία 10. Βάιλερ Μπέρμαν. Έχουμε μια συμβιβαστική τροπολογία εδώ. Υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 11. Χάρτογκ. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 13, τροπολογία 12, Βάιλερ Μπέρμαν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 14, τροπολογία 14, Βάιλερ Μπέρμαν, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13, Χάρτονγκ, είναι συμβατή με την τροπολογία 14 ως προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 15α, τροπολογία 15, Ανδρέασεν υπέρ, ανδρεα υπερ αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 16, τροπολογία 16, Χάρτον υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 17, τροπολογία 17, Ερενχάουζερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Τροπολογία 18. Χάρτονγκ. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 21. Τροπολογία 19 του κυρίου Χάρτονγκ. Έχουμε... Έχει ζητηθεί από το ΕΛΚΕ κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, μέχρι εκεί που λέει Facilitating Role. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα πρέπει να το ψηφίσουμε. Ωραία, δεύτερο τμήμα που λέει draws attention, το υπόλοιπο δηλαδή της παραγράφου υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές. Απορρίπτεται και αυτό. Ε, παράγραφος 25, τροπολογία 20. Αντρέασεν, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 27, τροπολογία 21 της κυρίας Αντρέσεν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 29, τροπολογία 23, Βάιλερ Μπέρμαν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22, Χάρτογκ, είναι συμβατή και μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 31α, νέα, τροπολογία 24, Ερενχάουζερ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 35, τροπολογία 25, Βάιλερ Μπέρμαν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 36, τροπολογία 26, Ερενχάουζερ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 45, ε, τροπολογία 27, Χάρτον, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 46, τροπολογία 28, Χάρτον, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 47, τροπολογία 29, πάλι Χάρτονγκ, Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, diplos de facto μέχρι financial management. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα να το ψήσουμε. Ναι, δεύτερο τμήμα. Regards this conduct. Το υπόλοιπο της παραγράφου. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και αυτό. Δεν είναι καλύτερη μέρα του κύριου Χάρτογκ σήμερα, μου φαίνεται. Παράγραφο 47α νέα, τροπολογία 30. Βάιλερ Μπέρμαν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 48α, 31 τροπολογία Χάρτογκ, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 48β της Επιτροπής Ανάπτυξης, τροπολογία 1. Ε, κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, διστάζω εδώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της Επιτροπής Ανάπτυξης αριθμός 1. Δεκατέσσερις έχουν ψηφίσει, κλείνει η ψηφοφορία. Αποτέλεσμα, 9 υπέρ, 4 ε, κατά. 13 ψήφισαν, άρα εγκρίνεται. Επόμενο τμήμα τρίτο υπέρ, κατά Εγκρίνεται. Παράγραφος 48 σε. Η δεύτερη τροπολογία της Αναπτυξιακής Επιτροπής, πάλι κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα στη τελευταία σελίδα, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 48 48Δ. Τρίτη τροπολογία της Αναπτυξιακής Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 48 Ε. Τέταρτη τροπολογία της ΔΕΒΕ, η χωριστά, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 48 σίγμα ταφ, εφ πέμπτη τροπολογία της ΔΕΒΕ, κατά τμήματα σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Δεν ξέρω, διστάζω. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Πέρα τη πληροφορία. Τι λέω υπέρ, λέει ο πρόεδρο, αφού είναι ηλεκτρονική. 8 υπέρ, 6 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές η ίδια πλειοψηφία όπως πριν εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Παράγραφο 48, ζήτα, ε, έκτη τροπολογία της ΔΕΒΕ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Ετελική τελική ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορία; Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είπαμε αποτέλεσμα 11 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Οπότε συγχαρητήρια κύριε Ρενχάουζερ για την τόσο καλή δουλειά που κάνετε και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ολομέλεια. Κύριε Γκρέσλερ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα, αυτό, μια μεγάλη ε, πολιτική ομάδα δεν είναι στι Βρυξέλλε. Δεν πάω αποδεχτούμε το τελευταίο. Η ομάδα μα είναι στη Μασαλία και έχει μερίδε μελέτη εκεί. Και έχει συνέδριο το ΕΛΚ λοιπόν και είναι όλοι στη Μασαλία. Ε, λοιπόν, ε, το ξέρανε σε κάποια ραδιοφωνική εκπομπή με την κυρία Τέισεν. Σας ακούσαμε, ναι, τηλεφωνικά από τη Βασιλεία. Δύο πράγματα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Έχετε μια πολύ καλή εικόνα του πώς είναι η ζωή μας έτσι. Ωραία, και να περάσουμε στις σημείο 4 λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στον ε, Επίτροπο, τον καλό να κάτσει λίγο πιο κοντά μου μάλιστα.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 Όπως ε, σας είπα και στις ανακοινώσεις του Προέδρου, θα δώσουμε κατόπιν αιτήματος των συντονιστών της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού το λόγο καταρχάς στον Επίτροπο Σεμέτα για να μας ε, επεξηγήσει την επιστολή που μας ε, απέστειλε για, για, το, για την απαλλαγή του Συμβουλίου ήταν δύσκολη η συζήτηση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν ο Επίτροπος μπορεί να μας διευκρινίσει. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη αυτής της Επιτροπής, μου απεστάλλει από τον Πρόεδρο στι 22 Νοεμβρίου μια επιστολή ζητώντα την άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα για τη σχέση μεταξύ του ε, ολοκληρώσεως των λογιστικών και των απαλλαγών όλων θεσμικών οργάνων και δεύτερον κατά πόσο ο δημοσιονομικό κανονισμό καλύπτει αυτά που θέλουμε. Ε, λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα και τα δύο θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι το κλείσιμο των λογαριασμών αυτό καθεαυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι η απαλλαγή θεωρείται δεδομένη. Το δεύτερο ερώτημά σας αφορά τις, πώς ταιριάζουν οι επιταγές συνθήκες με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι διατάξεις της συνθήκης, το άρθρο 319 πιο συγκεκριμένα, είναι σαφή όσον αφορά το θεσμικό όργανο προς το οποίο χορηγείται η απαλλαγή. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, άλλες διατάξεις της συνθήκης και του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπουν σαφώς την ε, συμμετοχή άλλων θεσμικών οργάνων και φορέων στη διαδικασία της απαλλαγής, κυρίως όσον αφορά τη συνέχεια πρέπει να δοθεί στο ψήφισμα της απαλλαγής. Αυτό έχει ερμηνευθεί ε, στη διαδικασία απαλλαγής επί δεκαετίας με τον τρόπο που γνωρίζουμε. Κατά άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διοικητική αυτονομία των θεσμικών οργάνων και η αρχή της ειλικρινούς αμοιβαίας συνεργασίας συνεπάγονται το ότι τα άλλα θεσμικά όργανα είναι υπεύθυνα και υπόλογα όσον αφορά τη διαχείριση του δικού τους ε, τμήματος του προϋπολογισμού. Το άρθρο 50 του Δημοσιονομικού Κανονισμού αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την εξουσία στα άλλα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν το δικό τους ε, τμήμα του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει την ευθύνη για την εκτέλεση αυτών των τμήματων του προπολογισμού και να ζητήσει την αλλαγή αυτών των συστημάτων που εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φρονεί λοιπόν ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργαστούν όσον αφορά τη δικασία απαλλαγή σεβόμενα τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης και τον σχετικό δευτερογενή, δευτερογενή νομοθεσία τη σχετική. Όπως είπα στην απάντησή μου, ελπίζουμε ότι ο διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δίδει νέα, θα, δοθεί, θα δώσει νέα όθηση συνεργασία στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία και σας διαβεβαιώνω εκ νέου ότι μπορείτε να βασιστείτε στους συνομιλητές από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αφοσιωμένοι σε αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Έχουν ζητήσει αρκετοί συνάδελφοι το λόγο και η Αγιάλα ζήτησε το λόγο που είναι η συγγήτρια. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Μάλιστα, η συγγήτρια λέει ότι θέλει να ακούσει πρώτα τους ε, ομιλητές, τους συναδέλφους. Από το ΕΛΚ, ποιος θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Χέλερ. Ευχαριστώ. Ε, ήθελα να ακούσω τυχόν σχόλια του ηλεκτρικού συνεδρίου. Θα ήθελα να σας ακούσουμε πριν μιλήσουμε εμείς. Εσείς τι θέλετε, δεν ξέρω. Uh, Αυτό που θα κάνουμε κατά αίτημα των ε, συντονιστών, ζητήσαμε τον από τον Επίτροπο να μας διευκρινίσει το γράμμα, την επιστολή για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Μετά θα δώσουμε το λόγο ε, στην συγκριτή για το θέμα της απαλλαγής του Συμβουλίου και τότε, όταν θα τα έχουμε τελειώσει όλα αυτά, θα δώσω το λόγο στο ελεκτικό συνέδριο στον Επίτροπο και μετά σε εσά ως εισηγητές. Αλλά ε, εντός του σημείου 4 ουσιαστικά έγινε μία μικρή αλλαγή της ατζέντα, την οποία και ανακοινώσαμε στην αρχή της συνδρίασης. Μάλιστα, δεν θα πάρω λοιπόν το λόγο τώρα. Ε, κύριε Γκάιερ, θέλετε το λόγο για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Ωραία, ναι. Και μετά η συγγήτρια, η κυρία Γιάλα Σέντερ. Συνάδελφοι, είναι αστείο μου ότι κανείς δεν θέλει να πει τίποτα για την επιστολή αυτή. Είναι, ναι, ναι, ναι, εσύ ήθελες, αλλά ήθελες να ακούσεις πρώτα να ακούσεις και την άλλη πλευρά. Να σας υπενθυμίσω. Αποφασίσαμε να μην δοθεί απαλλαγή μέσω αποχής στην Ολομέλεια και έτσι δημιουργήθηκε ένα θεσμικό ζήτημα οι σοσιαλδημοκράτες και εγώ προσωπικά ασφαλώς υποστηρίζουν την στάση της Επιτροπής ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να ε, είναι υπόλογο εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο για το θέμα του προπολογισμού. Αυτό είναι ασφαλώς θεωρητικά σωστό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι τυπικά και επίσημα δεν ε, ρυθμίζεται παρκώς. Μας αποκλείει το Συμβούλιο ουσιαστικά. διαβάσω την επιστολή του ε, ε, Επιτρόπου Σέμετα και αναφέρει ότι η τρέχουσα ερμηνεία τη δικαίου κτλ. Δεν μας προκαλεί έκπληξη αυτό. Ήταν και δική μας στάση άλλωστε αυτό. Θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε, θεωρώ, πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή. γιατί έχει αρχίσει μία κλιμάκωση. Δεν έχουμε κάτι άλλο στη διάθεσή μας. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και απόφαση του δικαστηρίου, γι' αυτό θα είμαι πολύ προσεκτικός, ότι υπάρχει δήλωση του Συμβουλίου ότι θέλουν να διαπραγματευτούν μαζί μας. Τώρα λοιπόν το ερώτημα που ανακύπτει είναι... Μπαρτ, ερώτησε σε επιστολή προς το Συμβούλιο το ποιο θα είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτό έχει διευκρινιστεί πλέον. Θα περάσουμε σε μια διαδικασία όπου εμείς ως Κοινοβουλευτική Ελεκτρική Αρχή είμαστε σύμφωνοι και αυτό θα δεσμεύσει το Συμβούλιο και θα πρέπει τώρα να κάτσουμε να σκεφτούμε υπό ποιου όρου θα ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει αυτέ. Αυτό είναι ακόμα επιτάπητο. Τι ξέρετε την επιστολή, αγαπητοί συνάδελφοι από το Συμβούλιο. Λάβαμε και σχετική επιστολή από την Προεδρία μάλιστα και οι συζητήσεις που διεξήχθησαν είναι ουσιαστικά και ερμηνεύονται με το εξή ερώτημα. Δεν ξέρουμε τι θέλετε, μα λέει το Συμβούλιο. Γιατί δεν είναι σαφές και διαφανές προς το Συμβούλιο πώς θέλουμε να διαμορφωθεί αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να ε, το τεθεί μια στοχοθέτηση, ίσω ένα μνημόνιο, δεν ξέρω. Ίσως θα πρέπει να γίνει κάποια α, τροποποίηση για να έχουμε και συμβατική ασφάλεια. Δεν αμφιβάλλει κανείς νομίζω ότι έχουμε δίκιο, αλλά στην πολιτική πάντα πρέπει να πάρει κανείς το δίκιο του κιόλας, όχι μόνο να έχει δίκιο. Ευχαριστώ, Γιέντς. Η κυρία Γκρέσλε και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Αγαπητέ συνάδελφε Γκάιερ, την εποχή του Δαρβίνη την έχουμε ξεπεράσει εδώ στην πολιτική. Έχουμε νομικές διαδικασίες και το ερώτημα στον Επίτροπο είναι κατά πόσον συμφωνεί με τη Συμβουλία. και μας απάντησε ο Επίτροπος ότι δεν συμφωνεί η Επιτροπή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω γιατί Τάλος αν ε, συμφωνούσε θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε από κοινού την απάλλαγη της Επιτροπής ε, και του Συμβουλίου. Άρα δεν είμαι απεσιόδεξη. Μπορούμε να διαχωρίσουμε τις διαδικασίες απαλλαγής. Αυτό νομίζω είναι καλή είδηση και για την Επιτροπή και αν είναι διαφορετική λοιπόν αυτή η αντιμετώπιση, θα δεθεί ξεχωριστά η απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα θα ρωτήσουμε τις ερωτήσεις που έχουμε να ρωτήσουμε στο Συμβούλιο και αν δεν απαντήσει, εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα ξαναξετάσουμε όλα αυτά, γιατί αυτό προβλέπει η νομοθεσία και είναι δικαίωμά μας. Και ας το ξαναοργανώσουμε το ζήτημα και να δούμε ποιος θα αντέξει πιο πολύ ποιος αντέξει και στο φως της δημοσιότητας. Γι' αυτό εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ξεχωριστή ειρήνη με το Συμβούλιο. Αυτά που έχουμε επιτάπητος παίζουν ρόλο στις δημοσιονομικές ε, διαπραγματεύσεις και είναι σαφές ότι το Συμβούλιο είναι υπόλογο προς εμάς. Αν το αμφι... αμφισβητεί αυτό, θα πρέπει να βγει και στη δημοσιότητα να το αμφισβητήσει. Αλλά αυτό δεν το αμφισβητεί ότι είναι υπόλογο. Αμφισβητεί ότι είναι υπόλογο σε θέματα προπολογισμού. Και γι' αυτό νομίζω ότι προχωρήσαμε στο θέμα αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου και τα υπόλοιπα νομίζω πρέπει να τα ρυθμίσουμε για την απαλλαγή με το 2010, ίσως και με βάση αυτά του 2009. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε την ίδια διαδικασία όπως το 2009. Δεν έχω ελπίδες ότι θα αλλάξει στάση το Συμβούλιο, αλλά επιτρέπε σε μέτα. Νομίζω ότι η κοινή γνώμη είναι πάντα νευρική με τα κόλπα που χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί το Συμβούλιο και τα χρησιμοποιεί και αύριο. Αμάν πια, τέλος. Η επιστολή του Συμβουλίου δεν αποτυπώνει την ε, άποψη της νομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν κατάλαβα καλά, επειδή διστάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι θραλέα μεν και συγχαρητήρια, αλλά δεν σύμφωνα με τον κύριο Γκάιερ, με τον συνάδελφο Γκάιερ, εγώ θα ήθελα να λάβουμε υπόψη και το ελεγκτικό συνέδριο. Το θέμα αυτό δεν είναι καινούριο. Το ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό. Το Συμβούλιο ε, θα συνεχίσει να κάνει κόλπα και το ζήτημα θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά. Και πιστεύω ε, αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλε, πάει η εποχή του Δερβίνου. Θα πρέπει, αν το Συμβούλιο, μάλλον αν εμείς που εκπροσωπούμε τους πολίτες, συγγνώμη, θα πρέπει να στραφούμε στο δικαστήριο. Και αν χάσουμε, χάσαμε. Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια μετά την πολιτική αυτή τοποθέτηση του Επιτρόπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κανείς άλλος πέρα από την εισηγήτρια. Η κυρία Γιάννα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι χτες υπήρξε αντίδραση από τις ομάδες από τις ομάδες μας σχετικά με το θέμα προτείνεται η ίδια τοποθέτηση όπως πέσει στον αφορά την απαλλαγή εμείς έχουμε διαφορετική τοποθέτηση θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο τον κύριο Σεμέτα για την απάντηση που έδωσε δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Επεξεργάζομαι το θέμα με την Επιτροπή και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη δυνατότητα διακυβέρνηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να βρούμε μια διέξοδο. Όταν ασχολούμαστε με αυτή τη διαφορά με τις σχέσεις των τριών θεσμικών οργάνων, ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει δεν θέλουμε απλώς να μας λέει κάποια πράγματα. Θέλουμε περισσότερο. Θέλουμε οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις σχέσεις του με το Συμβούλιο. Διότι έτσι ενισχύονται και τα τρία θεσμικά όργανα. Και με αυτό ακριβώς ασχολούμεθα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον Επίτροπο να το ξεκαθαρίσει αυτό. Έχουμε στην επιστολή που απεστάλλει από την νομική υπηρεσία μια καλή βάση. Όμως πρέπει να ε, μας δοθούν περισσότερα όσον αφορά την ενίσχυση της διακυβέρνησης και να ανταποκριθούμε και στις επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να λυθεί το θέμα της απαλλαγής με το Συμβούλιο. Έχοντας ακούσει τις διάφορες ομάδες, εγώ θα έλεγα ότι προτιμώ ως έχουν τα πράγματα και σχέση με το Συμβούλιο. Εγώ θα προτιμούσα, λέγω, να μην υπάρξει προσφυγή στο δικαστήριο. Δεν νομίζω ότι θα ήταν μια επιθετική δράση αν γινόταν κάτι τέτοιο. Είναι περισσότερο αντανακλαστική κίνηση θα έλεγα. Δεν θέλω όμως εμείς να βρεθούμε στην κατάσταση στην οποία θα είμαστε πιο αποδυναμωμένοι. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα το θέμα. Και υπάρχουν κάποιες πτυχές που είναι αρνητικές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών ίσως ακούσουμε άλλο ένα όχι, όπως προηγουμένως. Εγώ θέλω να εργαστώ επικοδομητικά όμως. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Διαφορετικά θα πρέπει να επαναληφθούν αυτά που έγιναν πέρσι. Όμως, αν εξακολουθούμε να λαμβάνουμε άσχημα αποτελέσματα, θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο θα έπρεπε να κάνουμε κάποια χειρονομία προς το Συμβούλιο, διότι ίσως να μην είναι σωστή κίνηση. Θα ήθελα να καταβάλει και άλλε προσπάθειε όμως ο Επίτροπος ο κύριος Σεμέτα και να αναγνωρίσει ότι κάνουμε καλή δουλειά, ότι κάνουμε περισσότερα πράγματα και ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε τα θεσμικά όργανα. Και, και κάνοντας το αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορέσει να συνεργαστεί μαζί μας εδώ. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους θεσμούς και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα, μα βοηθήσει και ο Επίτροπος, ο κ. Σεμέτα. Δεν θέλουμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση όπως πέρσι. Πριν προσφύγουμε στο δικαστήριο, νομίζω ότι θα πρέπει να στραφούμε προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν προσέφυγε στο δικαστήριο και υπάρχει μια δυνατότητα να δοθεί μια απάντηση και δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε αυτά που κάναμε κατά το παρελθόν γιατί ξέρουμε τα αποτελέσματα. Πρέπει απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας. Μάλιστα, την αποθέτηση τη εισηγήτρια σε ερώτηση προς και, στον, και προς τον Επίτροπο, αλλά έχω και τον κύριο Παλσίτη που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το θέμα μας απασχολεί επί μακρόν. Έχουν διεξαχθεί πολλές συζητήσεις. Δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε. Πολύ ευγενικά ο κύριος Επίτροπος ανέφερε κάποιες ε, λύσεις και είπε ε, τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Αυτή είναι η εντύπωση που σχημάτισα. Μετά σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάποιες αρμοδιότητες, κάποια καθήκοντα να εκπληρώσει και πιστεύω ότι οφείλουμε να πάρουμε μία απόφαση για τροποποίηση του κανονισμού. Έτσι θα ξεκαθαριζόταν τα πράγματα και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμορφωθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία. Και αν δεν το αρέσει αυτή η πρόταση του Συμβουλίου υπάρχουν και άλλες προτάσεις όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Πρόκειται περί έκφρασης πολιτικής βούλησης. Πρέπει να το κάνουμε αυτό και στη συζήτηση στην Επιτροπή δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να εκφράσουμε την πολιτική μας βούληση. Σας ευχαριστώ και πρώτα δώσω λοιπόν τον λόγο στον Επίτροπο. Η κυρία Γκρέσλε θέλει να παρέμβει εκ νέου. Ίσως ε, δεν ε, καταλαβαίνω τι γίνεται σήμερα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλουν οι συνάδελφοι στη τελική ανάλυση έχουμε κάποιες διαδικασίε. Δεδομένε. Έχουμε ένα κανονισμό, το δημοσιονομικό κανονισμό. Νομίζω ότι από τι διαδικασίες ως τώρα προκύπτει σαφέστατα ότι είναι υπόλογο το Συμβούλιο, αν και δεν το κάνει. Μπορούμε λοιπόν να τα γνωρίσουμε όλα αυτά ή μπορούμε να πάμε στο δικαστήριο. Όλα τα υπόλοιπα απλά δεν είναι εφαρμόσιμα. Εγώ θα ε- έλεγα να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε έως σήμερα. Να αποστείλει το ερωτηματολόγιο η εισηγήτρια, γιατί θα ήθελα να ξέρω τι άλλα περιλαμβάνονται για άλλε συμφωνίε με το Συμβούλιο. Για μένα δεν τίθεται θέμα. Είναι θέμα αρχή. Αυτό ο αμφότερο έλεγχο του προπολογισμού δεν τίθεται σαν αμφισβήτηση, γιατί εμεί είμαστε η αρχή απαλλαγή, χωρίς απαλλαγή. Αυτό ορίζεται από τη σύμβαση, από τη συνθήκη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να επιμείνω προς τον Επιτροπό να υπάρξει τοποθέτηση ε, της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής για την επιστολή του Συμβουλίου. Το νομική τοποθέτηση. Αυτό θέλω να καταρτιστεί. Χαίρομαι για τις απόψεις σας, μεν, αλλά η νομική τοποθέτηση είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε για τα επόμενα βήματα. Και κατά τα άλλα θα ήθελα να παρακαλέσω να μας αποσταλεί το σχέδιο ερωτηματολογίου, να μας δώσετε για τη σχετική προθεσμία, γιατί και εμείς θέλουμε ως ΕΛΚ να καταθέσουμε ερωτήσεις. Uh, θα θέλατε να ξαναπάρετε το λόγο? Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο, γιατί έχουν τεθεί ερωτήματα και από εσάς και από την κυρία Γκρέσλε. Και μετά μπορείτε να κάνετε, να ολοκληρώσετε ω εισηγήτρια το θέμα αυτό. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι αυτό το σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις συζητήσεις. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να βρουν μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία αποδεκτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την άποψή της και πρέπει να πω ότι αυτή η άποψη, παρόλο που είναι πολιτικής, ε, ε, δίνεται κατόπιν επαφής με την νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι απλώς μια πολιτική δήλωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο έλεγχος όλων των ε, θεσμικών οργάνων όταν μιλάμε για απαλλαγή και κάποιες ιδέες που ακούγονται να, ενταχθεί και το, να εμπλέκεται και το Συμβούλιο στην απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό θα έχει κάποιες συνέπειες. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνε αν δεν δύναται να έχει πλήρη, πλήρη δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης. και να εφαρμόζει και άλλες δράσεις που θα είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της ορθής οικονομικής διαχειρήσεως. Το θεωρούμε σημαντικότατο σημείο. Εγώ πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να δουν τις διατάξεις της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να δουν τι αναφέρεται. Εκεί ζητείται αμοιβαία ειλικρινή συνεργασία χρησιμοποιώντας τις διατάξεις της συνθήκης πιστεύω ότι θα βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση. Καταλαβαίνω την εξήγησή σας, αλλά ήταν, υπήρξε και μία σαφής ερώτηση από πλευρά τη κυρία Γκρέσλε. Λέτε ότι η πολιτική δήλωση αυτή μπορεί να Πρόκειται μάλλον για μια πολιτική δήλωση. Ασφαλώς πρόκειται για μια πολιτική δήλωση ενός επιτρόπου που βασίζεται επί μιας νομικής γνωμοδότησης. Αλλά κυρία Γκρέσλε νομίζω ότι η ρητά σας ρώτησε κατά πόσο μπορούμε να λάβουμε τη νομική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Επιτροπής. Είναι δυνατόν να τη λάβουμε. Τη βάση δηλαδή επί της οποίας προβαίνεται σε πολιτική δήλωση. Uh, Κοιτάξτε, δεν το θυμάμαι. Εγώ είπα ότι είναι πολιτική δήλωση που ετοιμάστηκε και συντονίστηκε με την νομική υπηρεσία. Ε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Δεν έχουμε μια ξεχωριστή νομική γνωμοδότηση επί του θέματος. Αυτές οι δηλώσεις που γίνονται στην επιστολή μου σχετικά με την ερμηνεία της νομοθεσίας έχουν γίνει κατόπιν συντονισμού, έχουν αναφερθεί κατόπιν συντονισμού συνεννοήσεως με την ε, νομική υπηρεσία της Επιτροπής. Ε, το προσπάθησα όπως και να έχει. Η κυρία Γκρέσλα και μετά η συγκεντριά. Στη Γερμανία λέμε ότι τα γραπτά μένουν. Έψαξα όλα μου τα χαρτιά, δεν βλέπω τίποτα γραπτό όμως. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρή αυτή η ιστορία. Δεν μπορώ να συστώ σε κάτι προφορικό. Θέλουμε γραπτά να μας πείτε ποιος δικαιούται τι. Γιατί τα γραπτά μένουν. Ο συνάδελφος Χατζημαρκάκης και μετά η συγγήτρια και μετά θα ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό πραγματικά γιατί έχουμε και άλλα σημαντικά ε, σημεία και έχουμε να ακούσουμε το ελεκτικό συνέδριο. Θα δώσω το λόγο και στον Επίτροπο. Βλέπω ότι επικρατεί ένας ενθουσιασμός. Θα δώσω το λόγο σε όλους. Ε, έχουμε την επιστολή του Επιτρόπου. Ο Επίτροπος αναφέρει στην επιστολή του ότι έχει συμφωνήσει με την νομική υπηρεσία της Επιτροπής. Άρα έχουμε κάτι γραπτό. Να σου δώσω, να σε δώσω την επιστολή μας. Έχει αποστείλει μια επιστολή ο Επιτροπός. Είναι διπλωματική η επιστολή, ίσως δυσνόητη, αλλά μας δείχνει δυνητικά δίκιο. Τελεία. Δεν είναι όμω απόλυτα σαφέ και 100% είναι πάρα πολύ διπλωματική η διατύπωση. Τώρα λοιπόν ρωτώ, μετά από την ερώτηση τη κυρία Γκρέσλε, καταλαβαίνω ότι δεν θα υπάρξει άλλη επιστολή, δεν πρέπει να, υπάρχει, να υπάρξει άλλη γνωμοτότηση Στην νομική υπηρεσία μεταξύ των θεσμικών οργάνων τα πράγματα είναι ω εξή. Αν δεν υπάρχει γνωμοτότηση, αυτή η αμφιλεγόμενο στοιχείο μεταξύ μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου θα πρέπει να επιληθεί εκεί που υπάρχει η αρμοδιότητα. Η Επιτροπή δεν συνεχίζει, δεν πάει παραπέρα, άρα στο δικαστήριο. Έχουμε την επιλογή να συνεχίσουμε όπως συνεχίζαμε ως τώρα. Αλλά είναι γεγονό ότι η κοινή γνώμη δεν ενδιαφέρεται και εκεί βασίζεται το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε όμω να συνεχίσουμε έτσι. Κατάλαβα τι είπε και η κυρία Αγιαλασέντρα και ο κύριο Μπαλτσίτης. Ότι θα πρέπει να περάσουμε πλέον στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση θα πρέπει να ζητήσουμε νομική γνωμοδότηση από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα πρέπει να ελέγξουμε τι διαδικασίε, τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μα, γιατί ο Επίτροπο μα το είπε ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να μα απαντήσει, δεν πρόκειται να μα δώσει οποιαδήποτε γραπτό στοιχείο. Ο κύριο Γκάιερ. Κανεί δεν είπε ότι πολύ απλά θα δώσουμε την απαλλαγή. Δεν πρόκειται να τα γνωρίσουμε όλα αυτά και ασφαλώς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία όπως ε, ως τώρα. Να είναι ήσυχη κυρία Γκρέσλε. Το θέμα είναι πώς θα επιλύσουμε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιλύσουμε αυτή την αντιπαράθεση τη θεσμική που έχει προκύψει με το Συμβούλιο και να την διευκρινίσουμε ε, κατά τη δική μας άποψη. Ε, συγχωρέστε με, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι μπορούμε κάποια ζητήματα να τα ξαναθέσουμε, θεωρώ. Καταρχά έχουμε τη δυνατότητα, το φροντίσαμε αυτό, έχουμε τη δυνατότητα στο νέο έτος, καταρχάς, για πρώτη φορά, να καλέσουμε την εκπροσώπηση, την αντιπροσωπεία της νέας Προεδρίας και να της θέσουμε τις ανησυχίες μας. Ήταν Η κυβέρνηση. Οι σκανδιναμικές κυβερνήσεις έχουν μία παράδοση μεγάλης διαφάνειας. Ενδεχομένω, λόγω παράδοσης, να ανταποκριθεί πιο πολύ η Προεδρία στις ανάγκες μας. Η Πολωνική Προεδρία συμπεριφέρθηκε τα αντίκεια, θεωρώ, αλλά ίσως να είχαν και άλλες προτεραιότητες. Μπορούμε να θέσουμε ένα κοινό κοινοβουλευτικό ερώτημα ως, ε, εκ μέρους της Επιτροπής, εκ μέρους των, ε, των ε, συντονιστών, μπορούμε να υποβάλουμε προφορικές ερωτήσεις και στην Ολομέλεια. Ούτε αυτό το έχουμε χρησιμοποιήσει ως δυνατότητα. Μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν συζητάμε ουσιαστικά και διαφωνούμε, απλά συζητούμε ποια εργαλεία έχουμε στην εργαλειοθήκη μας τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η πρότασή μου ήταν τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας να τα εξετάσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Goed, dan geef ik nu het woord aan de commissaris en dan... Ο Επίτροπος τώρα και μετά η συγκήτρια. Παρακαλώ, κύριε Επίτροπε. I just want to... Θέλω να επαναλάβω, να επιβεβαιώσω αυτά που είπα στην αρχή. Εσείς, ο πρόεδρος Επιτροπής σας μάλλον, ζήτησε γνωμοδότηση από αυτού παρουσιάσαμε γραπτός την άποψή μας με την υπογραφή μου. Την υποβάλαμε σε αυτή την Επιτροπή. Εξαρτάται τώρα από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο η εξέβρεση λύσης. Λύσεις στα πλαίσια των συνθήκων, όπου εκεί απαιτείται αμοιβαία ειλικρινής συνεργασία. Κάναμε αυτό που ζητήσατε. Και δεν είμαι σε θέση να δώσω κάτι παραπάνω. Εν συγκρίση με αυτό που ήδη έχω δώσει. Ε, Καλώς. Τέλος. Η συγκήτρια. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα του συναδέλφους. Νομίζω ότι η συζήτηση θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κοιτάξτε, αυτό που περιμένω είναι να έχουμε το ίδιο περιθώριο ελιγμών που είχε ο κύριος Ριβελίνη πέρυσι, που διαπραγματεύτηκε με το Συμβούλιο και κατάφερε ό,τι κατάφερε. Όπως είπε και ο κύριος Γκάγερ, λοιπόν, θα προσπαθήσω και ελπίζω, έχοντας εμπειρία από τη συναπόφαση, να καταφέρουμε κάποια στιγμή να προχωρήσουμε. Θα δούμε αν αυτό θα είναι εφικτό με τα μέσα που εσείς οι ίδιοι, κύριε Γκέσλερ αναφέρατε να πάμε και στο δικαστήριο ενδεχομένω. Αλλά αυτό βέβαια θα είναι το ίστατο εγχείρημα. Τώρα έρχομαι στον Επίτροπο για να είναι όλα ξεκάθαρα. Κύριε Σεμετά, καταλαβαίνω ότι εσείς την επιστολή σας την βασίσατε σε μια νομική γνωμοδότηση της νομοθετικής υπηρεσίας στην οποία απευθυνθήκατε. Όμω, επειδή εγώ δουλεύω και στι μεταφορές και έχουμε τη συναπόφαση καθημερινά μπροστά μα. συνηθίζω όταν το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο έχουμε κάποιες ιδέες αντιφατικές ή πάντων δεν συμφωνούμε μεταξύ μας. Τελικά η παντων δεν συμφωνουμε μεταξυ μα. έχει την υποχρέωση, είναι καθήκον της, οφείλει να βοηθήσει τα δύο θεσμικά όργανα να βρουν λύση. Και αυτό ζητάω από εσά. Εσείς λέτε στην επιστολή σας ότι η Επιτροπή θεωρεί επιθυμητό να συνεχιστεί ο μηχανισμός βάσει του οποίου το Κοινοβούλιο θα δώσει απαλλαγή και ε, απαιτεί από τα άλλα θεσμικά όργανα. Αχ, χτυπάει το κινητό μου, λέει η ομιλήτρια, το κλείνω. Έλεγα λοιπόν ότι απαιτείται διαφάνεια κτλ. Αυτό λοιπόν που εγώ σας ζητάω είναι εσείς να επιστρέψετε στις υπηρεσίες σας και να τους πείτε ότι πρέπει να μας βοηθήσουν, ότι πρέπει όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και εδώ, να βρούμε μέσα ιδέες, ε, τρόπους για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Πρέπει να μας βοηθήσετε. Το κοινοβούλιο μας σας το ζητά να μας βοηθήσετε. Εσείς λέτε ότι είναι επιθυμητό, ότι η Κομισιόν δηλαδή επιθυμεί να προχωρήσουμε για να δώσουμε την απαλλαγή, αλλά από εσά περιμένουμε φαντασία, δημιουργικότητα, να μας βοηθήσετε με τα κατάλληλα μέσα ώστε να βελτιωθεί η λογιστική διαδικασία και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να μην κλείσουμε δηλαδή εδώ το θέμα, αλλά από την πρόταση αυτή που μας ε, δώσατε με την επιστολή σας να συνεργαστούμε ώστε όπως ζητάει το κοινοβούλιο μας να μας βοηθήσετε και να βοηθήσετε και εμένα ως εισηγήτρια να προχωρήσω χρησιμοποιώντας νέα ή διαφορετικά μέσα ώστε τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο επαλήθευσης αλλά και μετά ενδεχομένως να μπορέσουμε να πάμε πιο πέρα με το Συμβούλιο και να αποφύγουμε το δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Οπότε το σημείο αυτό κλείνει εδώ. Μετά και κλεισμένο το θυρών, κατά πάσα πιθανότητα με τους συντονιστές δηλαδή, θα συζητήσουμε παρετέρω για αυτό το θέμα, ότι είχαμε να συζητήσουμε ανοιχτά, το συζητήσαμε. Θα δούμε με την εισηγήτρια στη συνέχεια και κλεισμένο το θυρών τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε. Και περνάμε τώρα στο πραγματικό σημείο 4 που είναι η απαλλαγή. Έχουμε εδώ πέρα μαζί μας από το ελεγκτικό συνέδριο την ε, κυρία Κάλιου Λάιτ, στην οποία και θα δώσω το λόγο. Παρακαλώ μέσα σε 8 λεπτά αν μπορείτε να έχετε ολοκληρώσει. Οπότε έχουμε εδώ και τον Επίτροπο που μπορεί να απαντήσει και στον εισηγητή φυσικά μετά θα δώσω το λόγο για ό,τι ερωτήσεις έχει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Κάλιου Λάιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε, αξιότιμα μέλη, κύριε Επίτροπε, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με την τήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή, την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2010. Να σας δώσω μία επισκόπηση των βασικών εξελίξεων όσον αφορά την παρουσίαση του κεφαλαίου 1 της ετησίας της Για την ετήσια έκθεση του 2010, η δομή τη ε, δήλωση εξοπιστία είναι διαφορετική. Όμω το περιεχόμενο δεν άλλαξε. Η ετήσια έκθεση εξακολουθεί να παρέχει μία άποψη όσον αφορά τον έλεγχο για την εξοπιστία των λογιστικών και των λογαριασμών και την τακτικό χαρακτήρα των συναλλαγών που υπόκειται των ε, λογαριασμών, δηλαδή ε, αναλήψη υποχρεώσεων και πληρωμέ και εισόδημα. Η γνωμοδότηση όσον αφορά τον τακτικό χαρακτήρα και των πληρωμών ε, είναι μόνο αντίθετη γνώμη. Εάν υπάρχει αιτιολογημένη άποψη, θα πρέπει να γίνει ποσοτικοποίηση του υπολογισμού των σφαλμάτων σύμφωνα με του νέου κανόνε περί ελέγχου. Γι' αυτό το δικαστήριο παρουσιάζει τη γενικό ποσοστό σφάλματο, πιθανού σφάλματο για τον εν γέννη. Πέραν αυτού, ε, για να παρασχεθούν πιο σαφείς ποσοτικοί δείκτες, τα ποσοστά για κάθε ομάδα πολιτικών δίδεται. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι ενώ αυτή αυτό είναι κάτι που αφορά τη γενική γνωμοδότηση, αλλά είναι η βάση μόνο για τα συμπεράσματα ανά ομάδα πολιτικών. Αυτά τα συμπεράσματα εξυπηρετούν για να δείξουν ποιοι είναι οι προβληματικοί τομείς ε, του προπολογισμού. Η μεθοδολογικό παράρτημα του κεφαλαίου 1 παραδίνει λεπτομερεί εξηγήσει σχετικά με το πώ υπολογίζει το ελεκτικό συνέδριο σύμφωνα με βασικέ στατιστικέ μεθόδου, του διάφορου ποσοτικού δείκτε και το, το ποσοστό ε, σφάλματο και το 90% περιθώριο εμπιστοσύνη. Η αιτήσια 6 του 2010 μα δίνει περισσότερε λεπτομέρειε για τι δύο μεγαλύτερε, για τη γεωργία και του φυσικού πόρου και τις σχετικές πολιτικές. Ενέργεια, μεταφορές και συνοχή μέσω δειγματοληπτικών στοιχείων για τις συναλλαγές. Θα ήθελα τώρα να στραφώ προς τα βασικά μηνύματα που βγαίνουν από την τύση έκθεση την φετινή, όπως ήδη παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο Καλτέρα τον... στις 10 Νοεμβρίου και στη σχετική συνεδρίαση που έλαβε χώρα. Το πρώτο βασικό μήνυμα είναι η εξοπιστία των λογαριασμών. Συνεπέρανε το συνέδριο για τέταρτο συναπτών έτος ότι οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δίνουν μια δίκαιη παρουσίαση πραγματική άποψη θα έλεγα της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων των διαφόρων ε, ροών των οικονομικών και των επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά όμως το ελεκτικό συνέδριο τόνισε και υπογράμμισε τι αλλαγέ όσον αφορά τη λογιστική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι πληρωμέ που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ταμεία που εφαρμόζουν διάφορα μέσα για οικονομική ε, διαχείριση. Το 2009 υπήρξε σημαντική αύξηση των πληρωμών που συμβάλλουν ε, στη δημιουργία και σύσταση τέτοιων ταμείων. Αυτέ οι πληρωμέ που έγιναν από τον πληθυσμό του 2000, το Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ενώση στα ταμεία, καταγράφονται σαν δαπάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ έχει καταγραφεί στα λογιστικά την εντύπωση ότι η χρήση αυτών των πληρωμών εδικαιολογείται σωστά από τους αποδέκτες της βοηθείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε έγκαιρη σωστή δράση για να διορθώσει τα υλικά προβλήματα όσον αφορά του προσωρινού λογαριασμού για το 2010 και επίση επανέλαβε και επιβεβαίωσε τα στοιχεία του 2009. Έλεγξε. Είδαμε ότι το ποσοστό των πληρωμών κάθε χρόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπό τη μορφή προκαταβολών που προχρηματοδοτούν το κόστο που ε, θα προκύψει αργότερα. Ε, το ποσοστό αυτών των προκαταβολών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του ενεστώτος δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, γι' αυτό υπάρχει σαφώς η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ε, του συστήματος υποβολής των οικονομικών στοιχείων, ώστε να αποκαλύπτονται σωστά οι κίνδυνοι που υπάρχουν για την οικονομική διαχείριση. Το δεύτερο μήνυμα της εκθέσεως αφορά τον τακτικό χαρακτήρα των συναλλαγών που είναι κάτω τα λογιστικά. Η έσοδα και δεσμεύσεις ε, ε, δεν είχαν σφάλματα, αλλά οι πληρωμέ επηρεάστηκαν από υλικά σφάλματα. Κατά 3,7% είναι το ποσοστό σφαλμάτων για δαπάνε γενικά τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αυτό το στοιχείο, το εκτιμόμενο ποσοστό σφαλμάτων, αντικατοπτρίζει τι συνέπειε των σφαλμάτων εκείνων που θεωρεί αρκετά σοβαρά το ελεκτικό συνέδριο για να τα ποσοτικοποιήσει. Αυτά τα ποσοτικοποιημένα σφάλματα συνδέονται με σοβαρέ παραβιάσει των κανόνων περί δημοσίων προμηθειών ε, και λανθασμένου υπολογισμού των κόστου που ε, ζητούνται τα κόστη αυτά να καλυφθούν από συγχρηματοδότηση από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ή λάθο δήλωση εκτάσεων από του γεωργούς. Λοιπόν, και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσωπικοποιηθεί. Σφάλματα που αναφέρονται μόνο στα στοιχεία περισυχνότητας και δίνουν κάποιες ενδείξεις τη δειγματοληψία που συμπεριλαμβάνει ποσοτικοποιημένα μη ποσοτικοποιημένα σφάλματα. Το 2010 οι πληρωμέ που δεν είχαν κανένα σφάλμα ήταν 64%. Ε, τρίτο βασικό μήνυμα της αιτήσης έκθεσης σχετίζεται με τις μεταφορές στην συνοχή ε, αυτή, αυτή την ομάδα. 7,7% είχαμε σε αυτή την ομάδα πολιτικών, μία αύξηση σε σχέση με το 2009. Αυτή η αύξηση υπεξηγεί τη μικρή αύξηση που σημειώσαμε στο γενικό επίπεδο ασφαλμάτων για το 2010 η αύξηση στο εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματος συνοδευόταν από μια αύξηση στη συχνότητα των σφαλμάτων. Σχεδόν οι μισές πληρωμές τώρα συμπεριλαμβάνανε σφάλματα. Επιπλέον, το ελεκτικό συνέδριο πίστωσε ότι οι αρχέ των κρατών μελών είχαν επαρκέ πληροφορίε διαθέσιμε, ούτω ώστε να έχουν εντοπίσει τα σφάλματα για 58% των πληρωμών που επηρεάστηκαν από ένα σφάλμα. Η αρνητική αλλαγή στον τομέα τη συνοχή θα πρέπει να δοθεί στα πλαίσια των όγκου δαπανών που περνούν από τα συστήματα. Αυξήθηκε από 23 δισεκατομμύρια στα 38 δις. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι στον τομέα της κοινή διαχείρισης έμεσα ελέγχει τα κράτη-μέλη το ελεκτικό συνέδριο όταν εξετάζει το κόστος των προγραμμάτων που χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ο έλεγχος οδηγεί στο να μπορούσαμε να συναγάγουμε συμπεράσματα αιτήσια όσον αφορά την ποιότητα των δαπανών για συγκεκριμένε πολιτικές, όπως η συνοχή. Το ελεκτικό συνέδριο δεν μπορεί να καταλήξει συμπέρασμα σχετικά τη διαχείριση των δαπανών συνοχής σε ένα δεδομένο κράτος μέλος τα πορίσματα για τι ομάδε πολιτικών είναι σχετικά σταθερά. Αυτό είναι το τέταρτο βασικό μήνυμα τη εκθέσεω του συνέδριου. 2,3% στη γεωργία και στου φυσικού πόρου είναι το ποσοστό σφάλματο, λίγο πιο πάνω από το υλικό κατόφλιο. Απ' την άλλη, φέτο το ελεκτικό συνέδριο έχει χτες πληροφορίε για να συμπεράνει ότι άμεσε πληρωμέ που διέπονται από το σύστημα ΔΕΑΚ είναι περίπου 70% των γεωργικών δαπανών και εκεί δεν είχαμε υλικά σφάλματα. Ενώ η ανάπτυξη υπαίθρου εξακολουθεί να δημιουργεί σφάλματα, να περιέχει σφάλματα. Για δύο ομάδε πολιτικών, έρευνα και άλλε εσωτερικέ πολιτικέ, η εξωτερική ενίσχυση, ανάπτυξη και διεύρυνση, ε, το ελεκτικό συνέδριο συνεπέρανε ότι οι πληρωμέ δεν είχαν υλικά σφάλματα. Παρ' όλα αυτά, Τόνισε το ρηκτικό Συνέδριο ότι η προσωρινή και τελική πληρωμή αυτών των ομάδων πολιτικών επηρεάστηκαν από διάφορα υλικά σφάλματα. Αυτό είναι σημαντικό διότι μόνο στην επιστροφή αξιώσεων για κόστο που αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον έχει γίνει, έχουν γίνει συμβαστοί κανόνε ή όχι. Και τέλο, όπω και σε προηγούμενα έτη, οι διοικητικέ δαπάνε παραμένουν ε, χωρί σφάλματα υλικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ε, ήταν η συντομευμένη ε, παρουσίαση της γραπτής, ε, του γραπτού κειμένου. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα. Κύριε Επίτροπε, εσείς να απαντήσετε. Thank you, Chair, honorable members. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή κυρία Καλιουλάιτ, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Θέλω να επικεντρωθώ στα κύρια σημεία που υπογράμμισε και το ελεκτικό συνέδριο, της πρωτοβουλίας μας δηλαδή προκειμένου να μειωθούν τα σφάλματα κυρίως στον τομέα της συνοχής και μετά να μιλήσω για τις επιπτώσεις στα επόμενα προγράμματα. Η εφαρμογή του προπολογισμού στους ε, τομείς όπου τον έλεγχο τον ε, έχουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη είναι ένα περίπλοκο θέμα. Δεν πιστεύω ότι ο σχεδιασμός του συστήματος υπό την τρέχουσα περίοδο είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι τα προβλήματα έχουν να κάνουν κυρίως με την μη ορθή εφαρμογή από τις εθνικές αρχές, μη ορθή εφαρμογή των κανόνων. Τα ευρήματα του ελεγκτικού συνεδρίου που λένε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δίνουν αρκετές πληροφορίες ώστε να εντοπίζονται κάποια τουλάχιστον σφάλματα, 58% δηλαδή των συναλλαγών που έχουν να κάνουν με τα σφάλματα, είναι κάτι που έχει κεντρική σημασία. Είναι απαράδεκτο να καταλήγουμε σε τέτοια λάθη. Μπορώ όμως να σας διασαφηνίσω ότι στα κράτη-μέλη έχω δώσει ευθύνε όταν παρενέβαινε στο ΕΚΟΦΗΝ την προηγούμενη εβδομάδα. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μπλοκάρει τις πληρωμές για όλα τα προγράμματα με επιφύλαξη και εκθέσεις που να δίνουν απαντήσεις στις ανησυχίες μας. Όλα αυτά ε, πάνε πέρα από τα προβλήματα τα οποία μέχρι τώρα αντιμετωπίσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 παρενέβη για 49 ERDF και για 14 πληρωμές ESF, του Κοινωνικού Ταμείου δηλαδή, ε, βάσει προθεσμιών. Και ενέκρινε και 6 αποφάσεις ε, παύσης. Η Επιτροπή συνεχίζει με την αυστηρή αυτή πολιτική της και το 2011. Για παράδειγμα, για τις πληρωμές ε, μπλοκ για την Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο σε 86 προγράμματα μέσα στο 2011 μέχρι τον Οκτώβριο και για την απασχόληση διέκοψε 16 πληρωμές και ενέκρινε μία απόφαση πάυσης. Από πλευράς πρόληψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να φέρει σε πέρας ελέγχους για προγράμματα που εγκυμονούν κινδύνους το 2011 και το 2012. Επιπλέον, η δημοσιευμένη ανάλυση των σφαλμάτων όσον αφορά την πολιτική συνοχή για τα έτη 2006 με 2009 δίνει μια καλή και λεπτομερή επισκόπηση που υπάρχουν κυρίως τα προγράμματα. Γίνεται και γεωγραφική ανάλυση που υπογραμμίζει τα ειδικά προγράμματα σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών. Παρόλο όμω, που περισσότερα από τα προγράμματα προχωράνε καλά, πρέπει να βασιστούμε στις ικανότητες που έχουμε εκεί όπου τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Η Επιτροπή λοιπόν επικεντρώνει την βοήθειά της στην ενίσχυση της εποπτείας και του ελέγχου σε αυτούς τους πιο αδύναμους παράγοντες προκειμένου να τους στηρίξει και να τους ξαναβάλει στο αυλάκι. Ε, μια άλλη προληπτική δράση έχει να κάνει με ε, υποχρεωτική ετήσια επισκόπηση των ε, διαχειριστικών αρχών στα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο ξεκίνησε από τα τέλη του 2010. Η Επιτροπή πιστεύει ότι αυτή η νέα υποχρέωση θα προσφέρει περισσότερες πληροφορίες και αξιοπιστία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρχές εφαρμόζουν την ε, πολιτική συνοχής μέσω διαφόρων προγράμματων για την τρέχουσα περίοδο. Τα διευθυντικά ταμεία τώρα και σχετικοί κανονισμοί τους για την περίοδο 2007-2013 έχουν τροποποιηθεί και έχουν απλοποιηθεί οι κανόνες. Τώρα υπάρχει η χρήση των καταποκοπήν ποσών και των μονάδων κόστους, όπως επίσης και των έμεσο κόστους, πάλι με βάση καταποκοπήν ποσά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές με παραδείγματα ε, καλών πρακτικών. Επιπλέον, η διαδικασία για την επιτάχυση των πληρωμών για διάφορα προγράμματα έχει προχωρήσει με αναθερμένα επίση προγράμματα και έχει απλοποιηθεί. Όλα αυτά τα μέτρα βοηθούν να απλοποιηθεί η εφαρμογή όλων των προγραμμάτων και ενισχύει την απορρόφηση των κονδυλίων. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στα μελλοντικά προγράμματα. Η Επιτροπή θέλει ε, το... η θέση της πολιτικής συνοχής για το 2013 να αποτελέσει μια βασική στρατηγική επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει τους στόχους του 2020. Οπότε, η επισκόπηση όλων των επιτευμάτων σχετικά με τους στόχους αυτούς θα αποτελέσει ένα κεντρικό στοιχείο της διαχείρισης των προγραμμάτων. Για να βελτιωθεί ακόμα καλύτερα η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για τις επόμενες γενιές προγραμμάτων να βασίζεται σε εταιρικέ σχέσεις, σε συμβάσεις κατά κάποιο τρόπο εντό εισαγωγικών με τα κράτη-μέλη. Αυτές οι εισαγωγικά συμβάσει θα επιτρέψουν τον έλεγχο της πρόοδου και θα διασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για να πετύχουμε τους στόχους μας που είναι κατά προτεραιότητα, όπως να ε, στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη και να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Επιτροπή επίσης προτείνει και ένα νέο ελεγκτικό πλαίσιο που να βασίζεται σε ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών που θα επιτρέψει να έχουμε περισσότερη αξιοπιστία όσον αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο που κάνουν οι εθνικές αρχές. Όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα, προβλέπονται και νέες διατάξεις που λένε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει ε, να αν αποτυχάνουν να εντοπίζουν και να διορθώνουν ε, τις ε, ατασταλίες πριν υποβάλουν για αποζημίωση ισχυρισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε χάνουν μέρος των πόρων. Μια άλλη, ένα άλλο μέσο που χρησιμοποιούμε για τη συνοχή ε, από την αρχή που αρχίσαμε τη συζήτηση μας το 2010, για την απαλλαγή του 2010 δηλαδή, έχει να κάνει με την χρήση των ε, ειδικών δημοσιονομικών μέσων. Αυτά τα μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για την αστική ανάπτυξη ή για άλλους σπόρους που έχουν να κάνουν ε, με την ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει τα κράτη-μέλη για τη σωστή εφαρμογή των λογαριασμών. Έχει ήδη ετοιμάσει μια, ένα σημείωμα κατευθυντηρίων γραμμών με τις βέλτιστες πρακτικές. Η Επιτροπή επίσης έχει προτείνει βελτίωση της τρέχουσας νομικής βάσης, κάτι το οποίο θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται από τις εθνικές αρχές. Η πρόταση αυτή θα υιοθετηθεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει πιο συγκεκριμένα να ε, κάνει τον έλεγχο των ειδικών δημοσιονομικών μέσων σε διάφορες χώρες μέλη. Για τους μελλοντικό κανονισμό η Επιτροπή έχει προτείνει ενισχυμένα ελεγκτικά συστήματα προκειμένου έγκαιρα να έχει πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση για την κατάσταση εφαρμογής. Ε, θα τελειώσω τώρα στο θέμα της απόδοσης λογαριασμών στα κράτη-μέλη. Το, ετήσιο, μάλλον το τρέχον σύστημα ε, το ετήσιο ε, δεν προβλέπει αρκετή αξιοπιστία όσον αφορά τη λειτουργία των ε, συστημάτων. Εκτός από ένα ή άλλες τέσσερις εθνικές δηλώσεις δεν δίνουν τις πληροφορίες που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε κάποια αλλαγή. Για να βασιστούμε στο άρθρο 317 της Συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στην πρότασή της για το δημοσιονομικό κανονισμό τις, δηλώσει, τις δηλώσεις μάλλον ετήσιες διαχείρισης, δηλώσεις οι οποίες πρέπει να υπογράφονται σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και θα ακολουθήσουν ό,τι έχουμε ε, χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα στον γεωργικό τομέα. Επίσης, η άποψη της ε, Επιτροπής είναι ότι εφόσον ε, τεθεί σε εφαρμογή σωστά το σύστημα αυτό, θα ενισχύσει την αξιοπιστία των χωρών μελών και θα διασφαλίσει και πολιτική απόδοση λογαριασμών για ένα σύστημα το οποίο φαίνεται να είναι αποτελεσματικό και να έχει νόημα. Πιστεύω ότι η απαλλαγή για το 2010 θα είναι μια επικοδομητική διαδικασία και μια χρήσιμη για όλους μας. Και για να τελειώσω, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και για την έκθεση ελέγχου όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό βασίζεται στο άρθρο 86.4. Πρώτον, η διακυβέρνηση. Εδώ επικεντρωνόμαστε στην καταπολέμηση της απάτης, στην διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και στην διαχείριση των εκτελεστικών υπηρεσιών. Και προκειμένου να καλύψουμε τις εντοπισμένες αδυναμίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει διάφορα μέτρα. Πρώτα απ' όλα, ενημέρωσε την στρατηγική της για την καταπολέμηση της απάτης, ε, προωθώντας μια στρατηγική καταπολέμηση τη απάτη σε κάθε υπηρεσία τη και νέους κανόνες ασφάλειας. Επίση, η Επιτροπή επί ευκαιρία αυτή θα ενισχύσει τι υπηρεσίε τη και του εκτελεστικού οργανισμούς για να υπάρχει συμμόρφωση απέναντι στην πολιτική ασφάλειας στην πληροφορική. Η Επιτροπή θεωρεί ότι χρειάζονται κάποιες αλλαγές μετά την υιοθέτηση της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού. Τώρα, για την πληροφορική συγκεκριμένα. Όσον αφορά τις ανάγκες οι οποίες έχουν εντοπιστεί στις ε, διάφορες επιστολές, η Επιτροπή ε, αποφασίζει μια νέα δομή για την διαχείριση της πληροφορικής. Κάτι το οποίο σημαίνει μείωση των ε, συστημάτων πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 2.500 σε 1.600 μέσα σε ένα χρόνο και καλύτερη ολοκλήρωση των συστημάτων πληροφορικής και άρα σημαντικές περικοπές. Τώρα, όσον αφορά τους, τη στρατηγική ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί προγράμματα δράση στου ε, τομεί των διαρθρωτικών ταμείων και τη έρευνα. Είμαι πεπισμένο ότι είναι ό,τι καλύτερο για να ανταποκριθούμε στι συστάσει που έχουν γίνει και για να προχωρήσουμε έγκαιρα στην εκτέλεση. Τέλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η απόδοση της IES για την ε, περίοδο του 2010 συμμορφώνεται στις διεθνείς προδιαγραφές για όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Έχει συνεισφέρει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συστημάτων της ελέγχου. Η Επιτροπή επίσης πιστεύει ότι οι υπηρεσίε δίνουν, ε, προσφέρουν κατάλληλα προγράμματα δράσης που ανταποκρίνονται στις αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί και διασφαλίζει ότι μέσω της ε, Audit Progress Committee θα φροντίσει για τον τακτικό έλεγχο και την αποτελεσματικότητα έγκαιρα στην εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Νομίζω ότι μας καλύψατε με το παραπάνω. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Και θα δώσω το λόγο στην εισηγητρία για να κάνει, στον εισηγητή για να κάνει μια πρώτη αξιολόγηση και να θέσει πλέον ερωτήσεις θα πρέπει να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τον Επίτροπο και τις υπηρεσίες του που μας έδωσαν την ομιλία γραπτά, γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο και ότι περιλαμβάνει πολλές, ε, πολλή προετοιμασία. Έχουμε και κάποιες ε, ερωτήσεις προς τον κύριο Πίλμπαξ και τον κύριο που θα έρθει σε μετέπειτα φάση. Ο κύριος Φιέλνερ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Ευχαριστώ κύριε Καλολάιτ. Ελπίζω να μην σπαταλήσατε όλη την ενέργειά σας και τα πυρομαχικά για τη συζήτηση επί των χαμένων σημείων του το Συμβούλιο και χρειαζόμαστε ενέργεια και εδώ. Τέτοια εποχή η λέξη πρόοδο είναι στην, καθημερι... στην ημερήσια διάταξη. Όλοι συνοψίζουν ε, τι έγινε το χρόνο και όλοι λένε σημειώσαμε πρόοδο. Ήμουν μέλο τη Επιτροπή αυτή από το 2004 και κάθε χρόνο αυτή την εποχή το μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να είναι σημειώνουμε πρόοδο, είμαστε στο σωστό δρόμο. Αν μετρήσει κανεί τι λέξει, προσπαθεί να εντοπίσει τι λέξει, βλέπει ότι όλο πιο συχνά χρησιμοποιούνται αυτέ οι λέξει προ το τέλο του χρόνου και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβεβαιώνει ότι οι τρέχουσες αδυναμίες θα διωθούν την επόμενη περίοδο και στον επόμενο κανονισμό. Και καταλαβαίνω αυτά που λέτε κύριε Επιτροπή, σα άκουσα και για το μέλλον αυτά που είπατε και μου αρέσουν, πρέπει να το παραδεχτώ. Ταυτοχρόνω όμως, στην αρχή της καριέρας μου σαν μέλο του Κοινοβουλίου, το έβρισκα, αυτά πιο καθησυχιστικά από ότι τώρα. Με τα χαράς μάθαινα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φέρει τελική ευθύνη για την εφαρμογή, την εκτέλεση του προπολογισμού, είχε την πεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μετά όμω, ακούγοντα την ίδια ταινία, την μαγνητοτενία, επί σειρά ετών, κατάλαβα το τρόπο με τον οποίο μιλάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει κάτι ανοιχτό. Κάθε χρόνο, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνει φανταστική πρόοδο, αλλά ποτέ δεν φτάνουμε εκεί που θέλουμε. Ποτέ δεν πετυχαίνουμε το στόχο και πάντα θέλουμε να πετύχουμε κάτι στο μέλλον, κάτι που είναι μπροστά μα συνέχεια και το κυνηγάμε. Και νομίζω ότι φέτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι σημειώνει η πρόοδο ακόμα και αν το ελεκτικό συνέδριο η κατάσταση παραμένει σταθερή σύμφωνα με αυτά που λέει το συνέδριο. Αλλιώ τα λέει το συνέδριο. Και παραθέτω. Το γενικό σύστημα ελέγχου και υποπτία, τα γενικά συστήματα αυτά είναι μόνο μερικώ αποτελεσματικά και οι πληρωμέ που βρίσκονται κάτω από του λογαριασμού μέχρι 31 Δεκεμβρίου εξακολουθούν να επηρεάζονται από υλικά σφάλματα. Τέλος παράθεσης. Το ότι μετατρέπει το μήνυμα του Ελεκτικού Συνεδρίου Ευρωπαϊκή Επιτροπή από σταθερό σε πρόοδο, νομίζω ότι είναι κάτι υπερβολικά αισιόδοξο. Κατά την άποψή μου, σταθερό δεν είναι πρόοδος. Και όπως προανέφερα, και θα επαναλάβω πιθανότατα πολλές φορές, το σταθερό δεν είναι καλό. Ας φύγουμε από τη σημειολογία τώρα. Και θα ήταν σε ευκαιρία να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδωσε μια απάντηση ε, που έδωσε απαντήσει γραπτό. Μα βοηθήσατε να ξεπεράσουμε τη σημειολογική συζήτηση για το πού ακριβώ βρισκόμαστε και ε, να μπούμε στην καρδιά του θέματο. Ε, θα ήθελα όμω να αναφέρω πέντε διαφορετικά σημεία ή θέματα. Πρώτα, έλεγχο και γενική διεύθυνση Ρίτζιο προετοιμαζόμενος για αυτή την ακρόαση, θα έλεγα ότι είσαστε το πιο σκληρό καρύδι για να προετοιμαστεί κανείς για να το μιλήσετε. Κύριε Σεμέτα, επίτροπε, Σεμέτα είσαστε επίτροπος υπεύθυνο για έλεγχο. Το μεγάλο ερώτημα που διερωτώ όταν ετοιμάζομαι, είσαστε υπεύθυνο για εκεί που βρισκόμαστε ή δεν είσαστε. Το θέμα του ελέγχου τώρα λοιπόν και της Γενικής Διευθύνσης Ρέτζιο. Θεωρείτε ότι είσαστε συνυπεύθυνο μαζί με τον Επίτροπο Χάν για την μείωση του ποσοστού σφάλματος του 7,7% στην πολιτική συνοχή. Πέρσι έγινε πολύ καλή συζήτηση, καταλήξαμε σε πολύ καλά συμπεράσματα για αναστολές και διακοπές. Και είπατε ότι αυξήθηκε ο αριθμός των διακοπών, είπατε μπλοκαρίστηκαν κάποια. Είπατε είχατε έξι αναστολές στην περιφερειακή πολιτική. Αυτά, τα, αυτές οι έξι περιπτώσεις ήταν από το κοινωνικό ταμείο. Το ε, ΦΕΟΓΚΑ όπου έχουμε το μεγάλο κομμάτι των προβλημάτων. Θα είναι πάνω από 7,7%. Είχαμε εκεί αναστολές. Ποιος είναι υπεύθυνο γι' αυτό έχετε κάποια επιρροή όσον αφορά τον τρόπο που η Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας, η για τις Περιφέρειες χειρίζεται τον προϋπολογισμό ή κάνουν ό,τι θέλουν στην DG Regio. Ήσαν υπεύθυνο για έλεγχο, έχετε λόγο όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούν, πώς τα χρησιμοποιούν. Έχετε λόγο, ε, έχει αρκετό βάρος. Ένα παράδειγμα. Υποτιθέστε ότι η DG Regio έχει εφεύρει κάτι που δίνει στα κράτη-μέλη μεγάλη ευελιξία. Και η DG Regio έχει καλές δυνατότητες να διανέμει τα χρήματα του προπολογισμού. Την άλλη, εσείς συμπεραίνετε ότι από πλευρά ελέγχου και του ποιος είναι υπόλογο, αυτό που εφήβραν είναι κάπως παρακινδυνευμένο. Εν τη αυτή περιπτώσει, ποια είναι η δική σας ευθύνη. Τι πιστεύετε. Ποια είναι η ευθύνη του Επιτρόπου που είναι υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Υπάρχει, είναι ξεκάθαρο ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Αυτή την πρόκληση αντιμετωπίζω εγώ όταν σα θέτω ερωτήματα. Ποιε είναι οι δικέ σα ευθύνε, πού ξεκινάνε οι ευθύνε σα, πού τελειώνει η ευθύνη σα. Αυτό το παράδειγμα με οδηγεί φυσιολογικά στη δεύτερη ερώτηση. Τα διάφορα μέσα για την ε, οικονομική διαχείριση. Financial engineering παίζει σημαντικό ρόλο στα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου του 2010 και καλωσορίζω την προσπάθεια που κατέβαλε το ελεκτικό συνέδριο στον τομέα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Στην ανάλυση του ελεκτικού συνεδρίου για την πολιτική συνοχή, μάλλον στην ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα σφάλματα στην πολιτική συνοχή, τα διάφορα μέσα οικονομικής ε, χειραγώγηση, αν θέλετε, financial engineering, ε, ε, αντιπροσωπεύουν μεγάλο κίνδυνο. Τι εννοείται με μεγάλο κίνδυνο. Τα έχει δηλώσει αυτά τα μέσα ότι είναι μεγάλο κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ξέρατε ότι είναι υψηλού κινδύνου ή είναι νέα έμπνευση κατά τη διάρκεια του, της φετινής εκτέλεσης. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί αυτά τα μέσα για την οικονομική ε, διαχείριση θα χρησιμοποιούνται πιο συχνά του χρόνου, αν είναι μέσα υψηλού κινδύνου. Το Financial Engineering. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις που θα θέλαμε γραπτές απαντήσεις, κυρίως για τα μέσα για το financial engineering. Στο πρώτο ήμιση ενός τέτοιου ερωτήματος απαντήσατε άριστα. Για το δεύτερο ήμιση όμως δεν απαντήσατε τόσο καλά. Ποιοι άλλοι ε, τομείς πολιτικής επηρεάζονται τα μέσα του financial engineering. Το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι υπάρχουν και άλλοι τομείς πολιτικής πέρα από τον προφανή της συνοχής και της αναπτύξεως της υπαίθρου. Βλέποντας την απάντησή σας, εξακολουθώ να βλέπω μόνο τη συνοχή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και είναι ένας τομέας όπου εμείς, ε, πώς να ε, αισθανόμαστε ότι οι έλεγχοι δεν λειτουργήσαν 100% και γι' αυτό είναι σημαντικό για μας να ξέρουμε επακριβώς πού χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα, αυτά τα εργαλεία. Μετά, τρίτον, αξιοπιστία όσον αφορά τη διαχείριση, πώς παρουσιάζει διαχείριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ που το τόνισε αυτό το τρεκτικό συνέδριο που αναφέρθηκε στη συνοπτική έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη γνωμοδότηση του εσωτερικού ελεγκτού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά μέσα ελέγχου αυτά, τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν εκ του σύνεγγυ από το Ελεκτικό Συνέδριο. Σαν Ευρωβουλευτέ, ξέρουμε ότι μπορούμε να του εμπιστευτούμε στο Ελεκτικό Συνέδριο. Και ανησυχώ κάπω διαβάζοντα πρώτα απ' όλα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποιε κατευθυντήρε γραμμέ για να εκτιμήσει το δικό τη ποσοστό σφαλμάτων Ίσως θα έπρεπε να πω ότι οι γενικοί διευθυντές μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και για να το πω ήπια και να εκτιμήσουν και με υπερβολική αισιοδοξία τα επίπεδα σπαλμάτων. Το συμπέρασμα του ελεκτικού συνεδρίου είναι ότι θα έπρεπε να υπήρχαν περισσότερε επιφυλάξει. Ποιο είναι το δικό σα συμπέρασμα, κύριε Σεμέτα. Δεύτερον, όσον αφορά τη γνωμοδότηση τη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είδα τα πορίσματα, δεν μπορώ να κρίνω κατά πόσο είναι χρήσιμα, αλλά μα λέει το ελεκτικό συνέδριο ότι το πεδίο εφαρμογή των νομοδοτήσεων είναι περιορισμένο στο, στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που όλοι γνωρίζουν ότι 90% των σφαλμάτων εντοπίζονται εκτό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, ποια είναι η άποψή σα, κύριε Σεμέτα, πόσο χρήσιμη είναι αυτή η γνωμοδότηση. Εγώ συμπεραίνω ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ότι χωρίς ουσιαστική επανεξέταση βάσει των πορισμάτων του ελεκτικού συνεδρίου είναι δύσκολο να δει κανείς την αξία που έχει εάν ε, του ξεφεύγουν αυτού του συστήματος το 90% των σφαλμάτων. Τέταρτον, η κυρία Καλουλάκη το ανέφερε αυτό επίσης, η αυξημένη χρήση της προχρηματοδότησης ή ο όρος προχρηματοδότηση ε, δεν ακούγεται σαν μια λέξη που θα μπορούσε να ενθουσιάσει έναν πολιτικό. Διαβάζοντας όμως ε, αυτά που λέει το ελεκτικό συνέδριο μου δημιουργήθηκε κάποια περιέργεια. Όλο και περισσότερο διακινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνοντας περισσότερους πόρους μέσω προχρηματοδότησης. Σαν δικαιολόγηση αυτών των πληρωμών έρχεται αργότερα, πολλές φορές πολύ αργότερα, πολλά χρόνια μετά. Και πιστεύω ότι το πρόγραμμα ε, διαβίου εκμάθηση είχε προχρηματοδότηση 100% αναπρόγραμμα πρόγραμμα και 93% όλων των πληρωμών που δόθηκαν το 2010 ήταν σε προκαταβολές. Αυτό είναι ε, απογοητευτικό, πώς να το πω. Πείτε μου κύριε Σεμέτα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναλάβει αυτό τον αυξημένο κίνδυνο και πώς μειώνεται αυτός ε, ο κίνδυνος. Ε, και διαρωτώ με. όταν το εξετάσατε το θέμα. Εξετάσατε το ενδεχόμενο το εξή. Λέτε, υψηλό επίπεδο συγχρηματοδότηση θα μείωνε το ποσοστό σφαλμάτων. Αυτό αναφέρει το ελεκτικό συνέδριο σε τομεί όπω εσωτερική πολιτική και εξωτερική βοήθεια. Το ποσοστό σφαλμάτων ήταν κάτι που ελήφθη υπόψη όταν κάνατε την ανάλυση της προχρηματοδότησης και κάτι εξής σημαντικό. Η οικονομική κρίση και ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μέτα, όπω προανέφερα, θέλω να καταλάβω το πώς εκτίθεται στου οικονομικού κινδύνους, χρηματοστατικού κινδύνους ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντα υπόψη την οικονομική χρηματοστατική κρίση που πλήττει τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή σα, πού εκτίθεται στους κινδύνους ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι μέτρα πήρατε για να μειώσετε αυτού του κινδύνου, αναφερόμενο στον πίνακα που μα δώσατε σε απάντηση του πρώτου ερωτήματό μα. Συνολικά εκρεμή ποσά την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι μέτρα έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χειριστεί τον οικονομικό κίνδυνο σε σχέση με τα εκρεμή αυτά ποσά ή δεν βλέπετε κάποιο κίνδυνο. Νομίζω ότι πολλοί από εμά είμαστε περίεργη. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του επομένου διημέρου. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω κινδυνεύει και αυτό τι επόμενε δύο μέρε. Ε, αυτά είναι τα ερωτήματα που έχω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σεγητά. Πολλές ερωτήσεις, πέντε συγκεκριμένα θέματα να προτείνω να μα απαντήσει ο Επίτροπος και μετά να εξετάσουμε ποιοι ζητούν άλλο το λόγο για τον πρώτο γύρο. Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε στα πέντε πρώτα θεματάκια που, έστει, που ρώτησε ο εισηγητής. Well, thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές ε, που έχουν να κάνουν με τις ευθύνες για τους ελέγχους. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια υπηρεσία ιστορικού ελέγχου, είναι μια κεντρική υπηρεσία και είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους στις υπηρεσίες. Έχουμε ένα σύστημα εσωτερικών ικανοτήτων για κάθε γενική διεύθυνση. Έχουμε ομάδες ελέγχου στις γενικέ διευθύνσεις. που διεξάγουν συγκεκριμένους ελέγχους στα κράτη-μέλη. Και φυσικά όλες αυτές οι δομές ε, σχετίζονται. Και για παράδειγμα, όταν γίνεται ιστορικός ε, ε, έλεγχος από τη σχετική υπηρεσία, Πέρσι έγινε έλεγχος και στον τομέα της συνοχής και προέκυψαν συγκεκριμένες συστάσεις από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου προς την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης για, να, για το τι θα έπρεπε να γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα των ελέγχων στο επίπεδο των κρατών μελών. Φυσικά, ο, ο συνάδελφος ε, Επιτροπός Χάν είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διαφορετικών ταμείων, όπως και ο Επιτροπός Άντερ, ο οποίος είναι υπεύθυνο και αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα παραστεί εδώ για την ακρόαση. Αυτή είναι η δομή λοιπόν που υπάρχει και που επιτρέπει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και έτσι μετά βάση συστάσεων λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις μέσω λοιπόν του εσωτερικού ελέγχου εφαρμόζονται και γενικές πολιτικές Επίσης τέθηκε το ερώτημα σε ό,τι αφορά τις αναστολές και τις διακοπές. Αληθεύει ότι έξι αναστολές έγιναν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αλλά πολλές διακοπές έγιναν επιπλέον στον τομέα του ERDF και κανονικά όταν γίνονται τέτοιες ε, διακοπές υπάρχει μια περίοδος 6 μηνών όπου οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να προβούν σε διορθώσεις στα συστήματα όπου έχουν εντοπιστεί ε, αδυναμίες και μετά τις διορθώσεις αυτές και οι, και οι διορθώσεις αυτές παρεμπιπτόντως υπόκεινται σε ελέγχους και αν η Γενική Διεύθυνση πιστεί ότι έχει βελτιωθεί το σύστημα δίνει εντολή για επανέναρξη των πληρωμών. Αν αυτό δεν ισχύει, συνεχίζεται η αναστολή των πληρωμών. Τώρα, για το, τα εργαλεία Financial Engineering. Και σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που προκύπτουν από τα μέσα αυτά. Φυσικά, όλοι θεωρώ ότι κατανοούμε ότι από μόνος του ο όρος Financial Engineering σημαίνει ότι εμπεριέχεται κάποιος κίνδυνος γιατί περιλαμβάνει ένα σύστημα εγγύησεων περιλαμβάνει χρηματοδότηση συγκεκριμένης μορφής μικρών επιχειρήσεων και τα μέσα αυτού του financial engineering ουσιαστικά έχουν ως σκοπό την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάφορες τομείς. Αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος μας, θεωρώ, να προωθηθούν οι μικρομεσαίες στα κράτη-μέλη. Ασφαλώς όλοι κατανοούμε ότι οι δραστηριότητε των νέων εταιριών, των νέων επιχειρήσεων, συνδέονται με κάποιους κινδύνους. Ασφαλώς, λοιπόν, θα πρέπει να λάβουμε κατάλληλα μέσα Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πιο καλούς συγκεκριμένους κατευθυντήριους κανόνες. Επίσης γίνονται συστάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν στα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι πρόκειται για ένα μέσο το οποίο ασφαλώς και αξίζει ε, την απόλυτη προσοχή μας. Γι' αυτό και γίνονται συγκεκριμένοι έλεγχοι. Ειδικά για τα μέσα του Financial Engineering. Εντάσσονται στο σύστημα χρηματοοικονομικής διαχείρισης για τομείς υψηλού κινδύνου και φροντίζουμε οι έλεγχοι να βασίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου. Άρα, οι επικίνδυνες αυτές δραστηριότητες υπόκεινται σε επιπλέον έλεγχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά οι επιφυλάξει του Γενικού Διευθυντή. Ξέρετε ότι σύμφωνα με το εφιστάμενο σύστημα, ο Γενικός Διευθυντής είναι εκείνο που αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη στην έκταση ετήσιας ε, δραστηριότητας και ο Γενικός Διευθυντής είναι αυτός ο οποίος ε, αξιολογεί όλους τους κινδύνους που ενέχονται σε όλους τους κλάδους της αρμοδιότητάς του, προκειμένου να προβεί ενδεχομένως σε επιφυλάξεις. Ε, εκτιμάται από το ελεκτικό συνέδριο ότι σε κάποιους τομείς χρειάζονται ίσως επιπρόσθετες επιφυλάξεις. Νομίζω λοιπόν ότι οι, γενικές, οι γενικοί διευθυντές ανέλησαν την γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου και προέβησαν σε ανάλογες αποφάσεις. Θα ληφθεί υπόψη ασφαλώς η γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ύστερα. Σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία των γνωμοδοτήσεων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη ότι ήταν η πρώτη φορά που καταρτίστηκε με τέτοια γνωμοδότηση. Αυτό αφενός. Κατά δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω άλλο θεσμικό όργανο με τόσο περιπλοκέ δομές που καταρτίζει τέτοιες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου. Ασφαλώς είναι περίπλοκο το ζήτημα, περίπλοκο το εγχείρημα. Αλλά το εγχείρημα αυτό μας επιτρέπει από τον πρώτο χρόνο κιόλα να πετύχουμε τον των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί συμμετείχαν στη φάση εφαρμογής των ελέγχων, όπου αυτό ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ποιότητα της τελικής γνωμοδότησης, χορηγώντας τις απαραίτητες πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό, θεωρώ. Γιατί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει βελτιωθεί σημαντικά. από την κοινή εργασία στο εγχείρημα αυτό. Φυσικά ομολογώ ότι το θέμα είναι η υπηρεσία ιστορικού ελέγχου να καταρτίζει την έκθεση αυτή για τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ το 90% των δραστηριοτήτων λαμβάνει η χώρα στα κρατημέλη. Συζητήσαμε το θέμα της συνολικής γνωμοδότησης στην Επιτροπή ε, Πρόοδου του Ελέγχου. Η Επιτροπή αυτή ζήτησε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου να εξετάσει τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και να σκεφτεί πώς πρόκειται να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, το οποίο δεν είναι ασφαλώς εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε καν στην εφαρμογή του λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμένους πόρους της υπηρεσίας εσωτερικού ε, ιστορικού ελέγχου. Δεν έχει δυνατότητα να διεξάγει ελέγχους και σε επίπεδο κρατών μελών. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος συντονισμός των ελέγχων που γίνεται από την υπηρεσία ιστορικού ελέγχου. Και θα πρέπει να χορηγούνται οι πληροφορίες από τους ε, ελέγχους που γίνονται σε επίπεδο κράτους μέλους. Και είναι σημαντικό θέμα και η ποιότητα των κρατικών, των εθνικών ελέγχων. Το ανέφερε αυτό και το ελληνικό συνέδριο. Δεν υπάρχει η ποιότητα αυτή των εθνικών ελέγχων. Αυτά λοιπόν τα θέματα βρίσκονται επιτάπητος και η υπηρεσία εσωτερικής, ε, εσωτερικού ελέγχου προσπαθεί να βελτιώσει την μεθοδολογία για την γνωμοδότηση. Ελπίζουμε ότι η επόμενη το δεύτερο έτος θα έχει καλύτερη ποιότητα. Τώρα, για την προχρηματοδότηση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την οικονομική κατάσταση, το οποίο και το πράξαμε σε ό,τι αφορά την προχρηματοδότηση. Η προχρηματοδότηση δεν έχει να κάνει με κάποιες ε, απόπειρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει το επίπεδο του σφάλματος. Αυτό δεν αληθεύει. Έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση, την οικονομική κρίση την οποία διανύουμε, το οποίο και σημαίνει ότι για πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν διαρθρωτικά ταμεία και τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ο μοναδικός τρόπος υποστήριξης της οικονομίας τους. Λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τα ελλείμματα που επικρατούν και την ανάγκη συγχρηματοδότησης των ε, πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, πολύ απλά δεν είναι δυνατή η απορρόφηση των ε, πόρων που διαθέτουν. Γι' αυτό λοιπόν ε, εισήχθη το σύστημα της προχρηματοδότησης και και πιο έντονα, ενδεχομένω να πρέπει ασφαλώς μάλλον θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στο σύστημα λαμβάνοντας υπόψη ότι η προχρηματοδότηση έχει καταστεί πλέον σημαντικό τμήμα της συνολικής χρηματοδότησης χωρίς όμως την δραστηριότητα αυτή Χωρίς την κίνηση αυτή, πολύ απλά πολλά κράτη-μέλη δεν θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που τους διατίθενται για να δώσουν μια όθηση στην οικονομία τους. Τελευταία ερώτηση για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού σε κινδύνους. Σας παρουσιάσαμε τις πληροφορίες που έχουμε για την δομή των πόρων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Φιλίπ Ταβέρν για να σχολιάσει το θέμα αυτό. Να το ζητήσω μάλλον να σχολιάσει το θέμα αυτό. Φυσικά επικρατούν κάποιες αβεβαιότητες και στον τομέα αυτό, αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν εκτίθεται. Υπάρχουν μακροπρόθεσμε, βραχυπρόθεσμε επενδύσει, για παράδειγμα, στη, στα κρατημέλη, τα, οι οποίες πρέπει να έχουν την ευρωπαϊκή υποστήριξη. Αλλά να ζητήσω από τον Φίλιπ Ταβέρν να επισέλθει λίγο πιο πολύ σε λεπτομέρειε. Ναι, να ζητήσουμε από τον κύριο Ταβέρνερ να απαντήσει την ερώτηση αυτή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα σας δώσω πρώτα μερικές συμπληρωματικές πληροφορίες για να απαντήσω στην ερώτηση αριθμός 1 καταρχήν. Δεν πρέπει να κάνουμε προσθέσεις και γι' αυτό και δεν τις κάναμε στο πίνακα, γιατί είναι για να, σαν να προσθέτουμε μήλα με αχλάδια. Είναι προφανές ότι η ερώτησή σας, έτσι όπως την καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, συνδέεται άμεσα με χρήματα τα οποία δίνει ο κοινοτικός προϋπολογισμός σε χώρες που βρίσκονται σε δυσκολίες. Ε, δεν σας μαθαίνω τίποτα καινούριο αν σας πω ότι αποφάσισε ένα κούρεμα 50% για την Ελλάδα το Συμβούλιο. Ε, πόσο από αυτό περιλαμβάνεται εδώ στον πίνακα. Στον πίνακα αυτόν έχουμε ένα ποσό το οποίο σήμερα, γιατί έχει να κάνει με τις 31 Δεκεμβρίου 2010, έτσι, δηλαδή τέλη Οκτωβρίου 2011, είναι 134 εκατομμύρια τα οποία βρίσκονται σε ταμείο εγγύσεων για τις εξωτερικές δράσεις και αλλού. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως, αν θέλετε, ο κίνδυνος για μας υπό το φως των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου είναι το μισό τελικά. Και επειδή εγώ ε, έχω αναλάβει με ο υπεύθυνο λογιστής για την Κομισιόν, μπορώ να σας πω ότι πέρα υπάρχει ένα impairment, δηλαδή μία συνεχούς βάσης μείωση. Και εννοείται ότι και υποχρώσεις κυμαίνονται. Αλλά το impairment είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι όταν πιστεύουμε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες λογιστικοί και όταν υπάρχουν τότε μπορούμε να έχουμε μία μόνιμη μείωση, impairment. Και αυτό ακριβώς κάνουμε τέλη 2011. Ποιο είναι το ακριβές ποσό δεν μπορώ να σας πω, γιατί στις 31 Δεκεμβρίου του 2011 θα μπορώ να σας το πω. Σήμερα όμως θα ήταν 50%. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους από το ελεγκτικό συνέδριο, όχι τα μέλη, τις υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Το έχουμε συζητήσει μαζί τους και με συμβούλους που είναι υπεύθυνοι για τη λογιστική, το τον πρόεδρο της Υψασφόρ κλπ. Τα θέματα αυτά είναι υπό έλεγχο. 67 εκατομμύρια είναι φυσικά κάτι περιορισμένο για την Κομισιόν. Τώρα, η άλλη μεγάλη κίνδυνη είναι οι δράσεις που θα έλεγα είναι back to back. Δηλαδή που έχουν να κάνουν με τα ισοζύγια πληρωμών για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης και μετά ερχόμαστε και στο μηχανισμό το EFSM. 2011 ξεκίνησαν βέβαια οι δράσεις, δεν ήταν το 2010, αλλά στο σημείο αριθμό 9 του Λεκτικού Συνεδρίου το έχετε, γιατί σας δίνει την παρουσίαση πώς είχε στις 27 Ιουλίου όταν υπογράφτηκαν οι λογαριασμοί. Μπορώ να σας δώσω και την κατάσταση πώς έχει σήμερα δεν υπάρχουν ιδιαίτερε δυσκολίε. Πρέπει να σα πω ότι η Ουγγαρία τα 2 δισεκατομμύρια που έπρεπε να δώσει τέλη Νοεμβρίου τα επέστρεψε χωρί πρόβλημα. Λέω χωρί πρόβλημα για μα, εννοείται. Πράγμα που σημαίνει ότι η πρώτη δοκιμή από τι πιστώσει ήταν επιτυχή. Τώρα, αν πάρετε τον πίνακα που επισυνάπτεται στο σημείο αριθμό 9, Ευχαρίστω αν θέλετε να βρεθούμε για να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως αν δείτε τον πίνακα αυτό βλέπετε ότι οι προθεσμίες είναι μεγάλες. Και αν κάθε μία, δηλαδή δεν είναι κοντά η μία στην άλλη, θέλω να πω ότι αν κάποια προθεσμία δεν τηρηθεί, δεν διακινδυνεύει ο προπολογισμό. Αν κάθε πιστωτής δεν πλήρωνε, κάτι το οποίο είναι πολύ απίθανο βέβαια, ο πρώτος πλήρωσε. Η επόμενη προθεσμία είναι μετά από μερικά χρόνια, δεν είναι τώρα αμέσω και φτάνουμε μέχρι το 2020 με τις προθεσμίες. Δεν λέω ότι υπάρχει μηδενικό κίνδυνος, θεωρητικά πάντα υπάρχει κίνδυνος, αλλά οι κίνδυνοι εντοπίζονται και τους παρακολουθούμε από κοντά. Ποια θα ήταν η διαδικασία κάποιο δεν πλήρωνε, ε, θα έπρεπε να παρέμβει η δημοσιονομική εγγύηση. Εννοείται, θα πρέπει να γίνει διορθωτικός προπολογισμό. Εννοείται και θα το κάνουμε σε μια πρώτη φάση στο εσωτερικό μας, μετά θα μπούμε στη δημοσιονομική διαδικασία αν χρειαστεί. Κατά τα άλλα στον πίνακα αυτών βλέπετε διάφορα πράγματα. Υπάρχει και ρευστό. Υπάρχουν και προβλέψεις όμως που συνδέονται με τον ίδιο το χαρακτήρα της οικονομικής κατάστασης. Υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται. Εγώ πάντως σας μίλησα για αυτό που φανάζει πιο πολύ, το πιο προφανές, το πιο προφανή κίνδυνο. Από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σας για να σας δώσω ό,τι άλλες εξηγήσεις επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ταβέρνα. Τώρα, να ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες, τους Σκιώδης δηλαδή, και ξεκινάω. Ποιος θέλει τον λόγο, ο κύριος Γκάιερ, Γκάιερ, ο κύριος Γκάιερ. Και μετά ο κύριος Χατζημαρκάκης και μετά ο κύριος Βόγγελ. Παρακαλώ κύριε Γκάιερ. Ε, κύριε Επίτροπε, σε μέτα δύο ερωτήσει έχω να σα κάνω. Η πρώτη για την προφορική μας ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Σας θέσαμε κάποιες ερωτήσεις ε, για τον τρέχοντα βαθμό ατασταλιών και τα στοιχεία για τις απάτες. Στες, κάναμε κάποιες ερωτήσεις για το πώς ε, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κριτική του ελεκτικού συνεδρίου σε σχέση με τα ανεπαρκή στοιχεία εκ μέρους των κρατών μελών για θέματα συνοχής. Όλα αυτά συνδέονται φυσικά. Αφενός είμαι ικανοποιημένος με τις απαντήσεις γιατί τονίζεται την ακρίβεια και την εντελέχεια με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βάλει στο σωστό δρόμο τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Από την άλλη το αποτέλεσμα είναι και πάλι απογοητευτικό παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε κάθε μέσο για να μειώσουμε το περιθώριο σφάλματος, βλέπουμε ότι αυξήθηκε εκ νέου. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Φιέλνερ, ο οποίος ρώτησε πώς σχετίζεται ο όρος πρόοδος που συχνά ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τέτοιες καταστάσεις. Λίγοι θεωρώ στην Επιτροπή μας θεωρούν το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επιληθεί στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είμαι κάπως διστακτικός σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κατά πόσον θα πετύχουμε το ποσοστό σφάλματος με διακή και βιώσιμο τρόπο να το μειώσουμε προκειμένου να φτάσουμε σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Συμφωνούμε εδώ στην Επιτροπή μας ότι θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαγραφεί μια τάση. Η τάση αυτή έχει διακοπεί εδώ και κάποια χρόνια. Ποιες είναι οι δικές σας ιδέες, κύριε Σεμέτα. Για την, για καμπύλη αυτή, για τις διακρινόμενες τάσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί και πάλι με το σωστό τρόπο. Δεν κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα θέλαμε να συζητήσουμε τις γενικές, τις αδρές γραμμές. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ποια είναι η γνώμη σας. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική συνέπεια όλων αυτών να είναι να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της η Επιτροπή να ανταποκριθεί. Και όλες οι εκθέσεις, όλα τα μέσα, όλα τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να βάλουν στο σωστό δρόμο τα κρατημέλη να εφαρμοστούν με άψογο τρόπο, αλλά να μην μπορούμε να ικανοποιηθούμε με το αποτέλεσμα. Είμαι πραγματικά άφωνος κάπως στην παρούσα φάση και θα θέλαμε να μας πείτε κι εσείς πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Δεύτερο ζήτημα από τις σημειώσεις μου. Το θέμα των τελωνίων δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, αλλά έχουμε, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν για να τεθεί το ερώτημα και μάλιστα να βάλουμε το δάχτυλο στην πληγή σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στις, ε, στα τελωνία των κρατών μελών. Ένα από τα σημαντικά ίδια μέσα που είχε ως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτώ λοιπόν, θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα των ε, στοιχείων που ζητούνται από τα κράτη-μέλη για, τα, για τις οριζόμενες ποσότητες το 2011 έχουν εκδοθεί καινούριε κατευθυντήριε γραμμέ για το τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η κατάσταση. Έχει καθαριστεί και έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ θα πρέπει να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα αυτά. Τι γίνεται ω προς το θέμα αυτό. Eh, Τώρα, ο Επίτροπος θα απαντήσει, αλλά Ναι, καλύτερα πρώτα να απαντήσει ο επίτροπο για να μην ε, ακούσουμε τι άλλε ερωτήσει, μήπω είναι για κάποιο άλλο θέμα. Uh, Όσον αφορά τα σταλίες και απάτες uh, που είναι το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης όπου θα συζητήσουμε την έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκεί εγώ θα παρουσιάσω κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για το θέμα. Η γενική μου αξιολόγηση από την έκθεση ποια είναι. Ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες συγκρίσεις. Συγκρίσεις μεταξύ ποσοστών σφαλμάτων που έχουν εντοπιστεί από το ελεκτικό συνέδριο, επίπεδο ατασταλιών, επίπεδο απατών και όταν πάρουμε τον τομέα της συνοχής, Φερρυπίν, το ελεκτικό συνέδριο κάνει μια εκτίμηση, ένα υπολογισμό σφαλμάτων. Επί τη βάση του χρησιμοποιημένου, του μοντέλου τους και της δηματοληψίας τους και φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα 7,7% για το 2010 οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τα κράτη-μέλη είναι συγκεκριμένα στοιχεία, δεν εκτιμήσεις, είναι στοιχεία που συλλέγουμε από τα κράτη-μέλη. Θεωρητικά λοιπόν το, η οροφή του επίπεδου σταλιών ίσως να είναι το ποσοστό σφάλματος που εκτιμάται από το ελεκτικό συνέδριο. Όσον αφορά το τομέα της συνοχής του 2010, το αναφερόμενο επίπεδα τασταλιών ήταν στο 3,15% στην συνοχή όπως σας είπα. εφαρμόσαμε πλήρως το σύστημα διαχείρισης ατασταλιών που επιτρέπει την αναφορά, ηλεκτρονική αναφορά των ατασταλιών με τρόπο φιλικό προς το χρήστη. Και αυτό είναι κάτι που αύξησε κατά πολύ την αναφερόμενη συμμόρφωση από τα κράτη-μέλη. και οι ατασταλίες επίσης εν γέννη θα μπορούσαν να εξηγηθούν από την εφαρμογή των νέων συστημάτων. Είναι καλό ταυτόχρονα ότι μπορούμε να εντοπίζουμε τις ατασταλίες, διότι κάθε ατασταλία οδηγεί σε συγκεκριμένη συνέχεια που δίδεται, δηλαδή ε, ανακτήσεις επίσης και τις σχετικές διαδικασίες. Αυτό καταδεικνύει ότι τα εισαγόμενα συστήματα αυτά αποδίδουν. Μας δίνουν κάποια αποτελέσματα ήδη. Όσον αφορά την τάση στο ποσοστό σφαλμάτων. Να πω ξεκάθαρα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το έτος 2010 ήταν το πρώτο έτος όπου το οικονομικό πλαίσιο 2007-2013 έφτασε στην πλήρη ταχύτητα. Άρα το επίπεδο πληρωμών, ε, τελικών πληρωμών προκαταβολών αυξήθηκαν δραματικά. Σχεδόν όλα τα προγράμματα ήδη ήταν καθοδόν υλοποίησεως. Παρά τούτο βλέπουμε ότι το επίπεδο σφαλμάτων που αξιολογήθηκε από το ελεκτικό συνέδριο στο ποσοστό του 7,7% είναι πολύ χαμηλότερο από την περίοδο 2008, 2007-2008, τα έτη 2007-2008. Άρα τα συστήματα μας έδειξαν ότι είναι σε θέση να εντοπίζουν τα προβλήματα και με κάνει συγκρατημένα αισιόδοξο. Πιστεύω ότι με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπουμε ή μάλλον που ήδη έχουν δρομολογηθεί μαζί με αυτά που προβλέπονται όλα αυτά θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε ε, ακολούθως και άλλες επιτυχίες στον τομέα. Έτσι ίσως απαντώ στο ερώτημά σας όσον αφορά τη μελλοντική πρόοδο. Αυτή η πρόοδος σχετίζεται πράγματι με σημαντική αύξηση των δράσεων όσον αφορά τους επιτοπίους ελέγχους. κάτι χρονοβόρο και που κοστίζει και σε ανθρώπινους πόρους, αλλά που θεωρούμε ότι αυτή η δράση είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία για να βελτιώσουμε την κατάσταση, βλέποντας επιτόπου τι συμβαίνει και τι μπορεί να βελτιωθεί. Έχουμε εντατικοποίησει την παροχή κατάρτισης, κυρίως στα κράτη-μέλη όπου βλέπουμε αλλαγές. Επί παραδείγματι, στους φορείς που χειρίζονται πόρους. Υπάρχουν κάποια προβλήματα όταν αλλάζει το προσωπικό και χρειάζεται εκ νέου κατάρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Και αυτό πρέπει να γίνεται συστηματικά. Έχουμε εκπονήσει ειδικά βασικό υλικό για την κατάρτιση που θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν καταφθάνει νέο προσωπικό και αρχίζει και εργάζεται σε συγκεκριμένο τομέα. Όσον αφορά τους τελωνιακούς δασμούς, είναι και αυτό κάτι που αναφέρεται στην έκθεση. μαζί με άλλους παραδοσιακούς ιδίους πόρους. Η, η Όλαφ, η ομάδα της Όλαφ προσέχει όλος ιδιαίτερο το θέμα. Πάντα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, αλλά τα τελευταία χρόνια εντοπίσαμε πολλές προσπάθειες αναταξινόμησης των αγαθών και υπηρεσιών, ούτως ώστε να επιτρέπεται καταβολή δασμών και αυτές οι δραστηριότητες εντοπίστηκαν από την Όλαφ και έγιναν τα δέοντα βήματα ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιστοφή χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο ερώτημα από ό,τι κατάλαβα αφορούσε τις αναγκαίες βελτιώσεις στους ε, ελέγχους στα κράτη-μέλη. Ναι, βέβαια παίρνουμε στα σοβαρά τα σχόλια, τα πορίσματα μάλλον του ελεκτικού συνεδρίου Δηλαδή λέει ότι τα κράτη -μέλη, στα κράτη-μέλη έλεγχη είναι εν μέρη αποτελεσματικά και ζήτησα ήδη από τις υπηρεσίες μου να ετοιμάσουν συγκεκριμένα σχέδια δράσεως για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασιζόμαστε κατά πολύ στο σύστημα των ελέγχων στους ελέγχους που παράγονται σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει να θέσουμε προτεραιότητα στην βελτίωση της καταστάσεως όσον αφορά το σύστημα ελέγχων των κρατών μελών. Ευχαριστώ, ο κύριος Χατζημαρκάκης. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι και στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Ίσως ο Επίτροπος θα μπορούσε, ίσως ο Πρόεδρος θα μπορούσε να μαζέψει, να μαδοποιεί τις ε, ερωτήσεις. Να συνεχίσω στην ερώτηση του κυρίου Γκάιερ για τα γενικά θέματα, για τις γενικές γραμμές, εντάξει, ε, συμφωνώ. Αλλά θα ήθελα με συγκεκριμένες ερωτήσεις να καταλάβουμε τις γενικές γραμμές. Σας ευχαριστούμε καταρχάς, ε, ε, κύριε Σεμέτα, για τις σαφείς δηλώσεις για τα κράτη-μέλη που κάνατε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ε, βλέπουμε ότι είναι πιο σκληρή η γραμμή έναντι των κρατών μελών και αυτό αποδίδει καρπούς και δικαίω. Αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στις δηλώσεις σας εδώ, αλλά και στις γραπτές σα απαντήσεις για τις διοικητικές σα δηλώσεις ε, τις υποστηρίζετε και λέτε ότι στην επόμενη προγραμματικό περίοδο θα είναι απαραίτητες και είπατε ότι σε διευθυντικό επίπεδο ε, διεξάγονται, αλλά θέλετε και πολιτική υποστήριξη. Πολύ ωραία. Αλλά πώς αντιδρούν τα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένη ερώτηση. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να υποχρεωθούν να δώσουν αποτελέσματα. Δεύτερο θέμα, το θέμα των διακοπών των πληρωμών που ανέφερε και ο συνάδελφος Φιέλνερ, αλλά είπε ότι γίνονται διακοπές αλλά όχι αναστολές σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής. Ερώτημα λοιπόν. Προγραμματίζετε ήδη, σχεδιάζετε το επόμενο επίπεδο της κλιμάκωσης, στο οποίο μπορείτε να προβείτε το ερωτώ γιατί μας υποβάλλεται και ένα έγγραφο εργασία όπου οι χώρες εκείνες όπου κυρίως παρουσιάζονται τα προβλήματα κατονομάζονται. Μία χώρα να αναφέρω γιατί επί σειρά ε, ετών, δεκαετιών εμφανίζεται η Ιταλία. Η Ιταλία και το ρωτώ συγκεκριμένα για να υποστηρίξει το ερώτημα του κυρίου Γκάιρ. Στην Ιταλία ξέρουμε ότι ε, ανήκει στις τρεις χώρες που ευθύνονται ε, για το 2 τρίτο των σφαλμάτων. Ξέρουν οι αρχές ακριβώς τι γίνεται. Και βλέπουμε ότι παρόλα αυτά τέσσερις υπάλληλοι δεν τηρούν τις ε, κανόνες. Εξακολουθεί ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις πληρωμές. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί, γιατί δεν... δεν μπορούμε να προβούμε όχι σε διακοπές των πληρωμών, σε αναστολή το πληρωμών να πούμε ότι κοιτάξτε Ιταλοί, δεν σα τα δίνουμε τα λεφτά αυτά. Νομίζω ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί σε κάποια φάση θα πρέπει να περάσουμε και στην επόμενη φάση της κλιμάκωσης, στην καταγγελία της χώρας αυτής. Το ξέρει ο αρμόδιος επίτροπος ότι οι αρχές γνωρίζουν μέν τους κανόνες, αλλά αρνούνται να τους εφαρμόσουν. Θέλω μια σαφή απάντηση. Τρίτη ερώτηση. Για την ε, την ανάκτηση των ποσών. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Το επιβεβαιώσατε αυτό και στις αιτήσει εκτέσεις σας. Τι θα κάνουμε με τα χρήματα αυτά. Ένα φωτικό παράδειγμα να αναφέρω. Από τον τομέα της αγροτικής ε, πολιτικής. Ο σχετικός επιτρόπος στις 14 Οκτωβρίου 2011 σε δήλωσή του δεν είπε μόνο πόσα χρήματα ε, ζήτησε 240 εκατομμύρια ευρώ αλλά ανέφερε και ποιες χώρες πλήττονται. Αυτό είναι πολύ καλό και διαφανές, αλλά απευθύνεται μόνο στη γεωργική πολιτική. Ερωτώ, το έχουμε συζητήσει και σε άλλο επίπεδο. Γιατί δεν λειτουργούν αυτά σε επίπεδο πολιτικής συνοχής, όπου ε, χορηγούνται τα μέσα και πληρώνονται και διαπιστώνονται ότι έχει γίνει λάθος, να ζητείτε ανάκτηση και να υπάρχει άμεσα αναστολή των πληρωμών. Και πώς θα βρούμε τα 3,5 δισεκατομμύρια που μας χρωστάει η Ισπανία, για παράδειγμα. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Θα ακολουθήσω τις ε, προτάσεις σας και θα οματοποιήσω τις ερωτήσεις ε, Βόγκεν και μετά Γκρέσλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω τρία συγκεκριμένα σημεία που θέλω να θίξω. Πρώτα απ' όλα, βάσει αυτού που είπε ο τελευταίος Το τελευταίο θέμα που αφορά τη διακοπή και αναστολή των πληρωμών. Από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ένα σύστημα. Σύστημα για διακοπή και αναστολή των πληρωμών. Το ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολίτες πώς ανακαλύπτουν για τις διακοπές. Επί γνωρίζω ότι κατά πρόσφατο παρελθόν πληρωμέ διακόπησαν προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Κανεί δεν το γνώριζε. Δεν ξέρουμε για ποιου λόγου. Δεν ξέραμε τίποτα εκ των προτέρων κατά τη διάρκεια τη διακοπή. Ερώτημα. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι πληροφορίε που σχετίζονται με τις διακοπές, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει περί αυτών και να ξέρει και του λόγου για τη διακοπή. Δεύτερο, απορρόφηση, ποσοστά απορρόφησης που αναφέρονται, αναφέρθηκα στην αρχική σα παρέμβαση. Μεγάλο πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει όχι στην Ουαλία να προσθέσω, αλλά στην Αγγλία πιο συγκεκριμένα. Και όσον αφορά την έλλειψη διαθεσίμων πόρων για διαθετικά ταμεία, προγράμματα διαθετικών ταμείων. Και αυτό σχετίζεται με τις περικοπές των δημοσίων δαπανών, βέβαια. Πείτε μας, θεωρείτε ότι υπάρχει και αλλού αυτή η τάση στην Ευρώπη. Ε, ποιες χώρες έχουν πρόβλημα όσον αφορά να βρουν την κατάλληλη χρηματοδότηση για την διάθεση των διαθωτικών πόρων από τα ταμεία και αν υπάρχει πρόβλημα τι υποτίθεστε να κάνετε. Τέλος, τα νέα χρηματοστικά εργαλεία που ανέφερε ο εισηγητής στη δική του παρέμβαση. Πρόσφατα είδα το Ταμείο Τζέρεμι που έχει σαν στόχο δανειοδότηση μικρομεσών επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβητεί από ό,τι ξέρω τη νομιμότητα κάποιων πληρωμών ε, για λόγους σχετίζονται με κρατικές ενισχύσεις. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Το γνωρίζετε. Αν το γνωρίζετε, τι πρόκειται να κάνετε. Διότι όπω είπε ο συζητητή, αυτά τα ανέχουμε μέσα μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικά στο μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Να επανέλθω στο θέμα τη χρέωση των κρατών μελών και του πόσο αξιόπιστε είναι οι χρηματοπιστωτικές διορθώσεις. Θα ήθελα να μου πείτε πως χώρες όπως ε, η Ισπανία και η Ελλάδα πρέπει να κάνουν τις διορθώσεις. Καταρχάς, ε, γιατί επίπεδο διορθώσεων μιλάμε και στον αγροτικό τομέα και στο διαφορετικό τομέα και σε ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία είναι οι βασικές χώρες. γιατί σε κάποια φάση δεν θα μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά με οικονομικές διορθώσεις. Θα θέλαμε επίσης μία, ένα πίνακα. Σε ό,τι αφορά τα ποσά αυτά και τις διακοπές αυτές στις χώρες. Θα θέλαμε ένα follow-up της κατάστασης. Goed, zijn er Καλώς, άλλος κανείς θέλει το λόγο. Θα έλεγα να δώσω το λόγο τώρα σε όποιον θέλει, να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις. Ε, μια ερώτηση ακόμα, παρακαλώ. Τώρα. Ναι, και ευχαριστώ. Συγγνώμη που μόλις έφτασα, είχα μια άλλη συνεδρίαση. Θέλω μια διευκρίνηση σχετικά με μια γραπτή ερώτηση. Την αριθμό 46. Η ερώτηση είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται την ευθύνη για την απαλλαγή του Συμβουλίου από μόνη της. Και έχω μια λεπτομερή απάντηση. Όμως, η... μπορείτε να συνοψίσετε με ένα όχι. Αυτό απαντάτε βασικά. Όσον αφορά την ερώτησή σας, λέει ο Πρόεδρος, μιλήσαμε επί τρία τέταρτα στην αρχή της συνεδρίασης. Εντάξει. Θα επανέλθουμε εξάλλου και στους συντονιστές. Εσείς είσαστε συντονιστή, οπότε θα τα ξανακούσετε και εκεί. Άλλη ερώτηση? Όχι? Καλώς. Ο Επίτροπος τότε, ενδεχομένως και το ελεγκτικό συνέδριο, εφόσον επιθυμείτε, και σίγουρα και στον εισηγητή, έτσι, ο οποίος μπορεί να επανέλθει σχετικά με όλα. Παρακαλώ. Ο κύριος Σεμέτα. Ήταν μια ομάδα ερωτήσεων που αφορούσε αναστολή και διακοπή πληρωμών. Όπως προανέφερα, δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά τα μέσα και όλες οι διακοπές που λαμβάνουν χώρα ακολουθούνται παρακολουθούνται μάλλον από τους ελεγκτές μας. Δεν είναι απλώς κάτι γραφειοκρατικό, παρακολουθούν πράγματι κατά πόσο έγιναν ιδέουσες βελτιώσεις για να ξαναγίνουν οι πληρωμές, να ξαναρχίσουν οι πληρωμές. Και είναι αρκετά σαφείς οι κανόνες. Αν υπάρξει βελτίωση μετά την διακοπή, και τα αίτια της διακοπής πάβουν να υπάρχουν, τότε ξαναρχίζει η πληρωμή. Και δεν οδηγούμε θα αναστολή των πληρωμών. Αυτή είναι η περίπτωση που θα εξηγήσει η συνάδελφος Χάν. Που θα το συζητήσει μαζί σας. Και να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Και όπως και ο Επίτροπος Άντερς όσον αφορά τις χώρες Ιταλία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Πρέπει να ασχολούμεθα με όλα τα κράτη-μέλη στο ισχύον νομικό πλαίσιο και το υπάρχον νομικό πλαίσιο προβλέπει τα προαναφερθέντα μέσα. Βέβαια, όταν εντοπίζουμε νέα προβλήματα σε συγκεκριμένα προγράμματα ή σε συγκεκριμένους τομείς, είμαστε πολύ προσεκτικοί και κάνουμε τα δέοντα. Διακοπές, πάυση πληρωμών, διακοπή πληρωμών. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε όμως όλες τις πληρωμές προς ένα κράτος μέλος, διότι δεν είναι κάτι που προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής. Όσον αφορά τις ανακτήσεις, μια ερώτηση του κυρίου Χατζημαρκάκη και της κυρίας Γκρέσλε. Το παράρτημα των ετήσιων λογαριασμών παρουσιάζει Στο σημείο 6, στο σημείο 6 παρουσιάζεται μια κατανομή των οικονομικών διορθώσεων και των ανακτήσεων κατά κράτος μέλος. Βλέπετε συγκεκριμένα ποσά βέβαια οι διορθώσεις που αποφασίζονται οι μεγάλες, για τις μεγάλες διορθώσεις που αποφασίζονται χρειάζεται χρόνος για τις ανακτήσεις για να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν. Για χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, ή άλλες χώρες, αν υπάρχει πρόβλημα, αν τα χρήματα δαπανώνται παράτυπα ή εντοπίζονται σφάλματα από το ελεκτικό συνέδριο ή από τους δικούς μας ελέγχους, παρά την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά τα κράτη-μέλη, πρέπει να ανακτήσουμε αυτά τα ποσά. Και θα το κάνουμε, αυτό είναι σίγουρο. για τη διακοπή και αναστολή πληρωμών κάτι ξέχασα και την δημοσιότητα, την γνωστοποίηση αυτών. Υποθέτω ότι τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν όταν παίρνουν το σημείο με την ανακοίνωση διακοπής πληρωμών. μπορούμε να λάβουμε και υπόψη και αν υπάρχουν κάποια, να εξετάσουμε αν υπάρχουν προβλήματα ευαισθητοποίηση σε κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά το θέμα αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση, να ενημερώνεται το κοινό, να βελτιωθεί εν γέννη η κατάσταση για την γνώση για το θέμα των διακοπών και αναστολών. στο κείμενο το κείμενο αυτό για τους λογαριασμούς μας είναι δημοσιόγραφο. Το έντυπο αυτό. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν και αυτά να πάνε στη χώρα τους και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο έντυπο και που παρουσιάζονται κατά κράτο μέλο και να χρησιμοποιήσουν το έντυπο αυτό για να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτά τα κράτη-μέλη. Υπήρξε και ένα ερώτημα για το Τζέρεμι και τα μέσα χρηματοστητικής μηχανικής financial engineering και το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Εν τη αυτή περιπτώση εφαρμόζονται γενικοί κανόνες. Και η οδήποτε είδος κρατικής ενίσχυσης, κρατικής βοήθειας ε, τελεί υπό την επιφύλαξη εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν εντάσσεται στα κατάλληλα πλαίσια, όρια ανεξάρτητα τον τρόπο χρηματοδότησης. Αν ξεπερνά το όριο, η χρηματοδότηση, και είναι... Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να εγκρίνεται η κρατική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αδίποτε κρατική ενίσχυση σχετίζεται με κίνδυνο. Μείωση ανταγωνισμού, Φερρυπίν. Και εφαρμόζει αυστηρότατη πολιτική περί ανταγωνισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς προσεκτικότατα τις κρατικές ενισχύσεις. Πιθανότατα απάντησα σε όλες τις τεθήσεις ερωτήσεις μέχρι τώρα. Α, ναι, όσον αφορά το Συμβούλιο, ήταν το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε ε, λεπτομερέστατα. Τώρα Ε, θέλετε εσεί να παρέμβετε τώρα κύριε Σιγητά. Εγώ σκεφτόμουν να δώσω πρώτα το λόγο στο λεπτικό συνέδριο στην κυρία Γιαγιουλάιτε και μετά, αν ήθελε να σχολιάσει δηλαδή, πάνω σε αυτά που ακούστηκαν και μετά να δώσω σε εσά το λόγο. Ναι. Αλλά έχω και κάτι στο οποίο θα μπορούσε εκείνη να απαντήσει για να μην ε, επανέρχεται. Εντάξει, τότε σας ακούμε. Ναι, θα είμαι σύντομο τώρα και μετά θα επανέλθω. Λοιπόν, όσον αφορά τι επιφυλάξει στι οποίε αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν κατάλαβα από αυτά που λέτε, όσον αφορά τις επιφυλάξεις, ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη, διαβάζει τι λέει το ελεκτικό συνέδριο και μετά το λαμβάνει υπόψη. Και έτσι μπορούμε να ελπίζουμε σε πρόοδο ότι θα είναι καλύτερα δηλαδή τα πράγματα στο μέλλον. Αλλά αναρωτιέμαι, είναι η πρώτη χρονιά που το λεκτικό συνέδριο το αναφέρει με επιφυλάξει. Γιατί αν είναι η πρώτη χρονιά, τότε εντάξει. Δεύτερον, με κάθε σεβασμό, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κοιτάει μόνο τις γενικές διευθύνσεις. Νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε στο θέμα των επιφυλάξεων και τις ευθύνες των επιτρόπων. Οι επιφυλάξεις εμφανίζονται το συνθετικό κείμενο, το οποίο το εγκρίνει το σώμα των επιτρόπων. Οπότε θα έπρεπε παντού να είναι σωστά τα πράγματα. Και αν το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερε επιφυλάξει, τότε ελπίζω ότι έχετε δίκιο ότι οι γενικέ διευθύνσει θα ακούνε το ελεκτικό συνέδριο, αλλά θέλω να ξέρω, το έχει ξαναπεί και προηγούμενε χρονιέ αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Αλλιώ πρέπει να φροντίσετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να επιβάλλετε να γίνεται αυτό. Εσείς με κάποιο τρόπο. Το λέω πριν ακριβώς απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο, ώστε να το συμπεριλάβει στην απάντησή της και αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τις επιφυλάξεις για τις αιτήσεις εκθέσεις δραστηριοτήτων, από όταν υπήρχαν, είπαμε ότι υπήρχαν επιφυλάξεις που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται, αλλά έλειπαν. Και ελπίζω ότι αυτές οι επιφυλάξεις να μην βασίζονται μόνο επί της δουλειάς που έκανε το ελεκτικό συνέδριο, διότι όταν γίνονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσανατολιστεί από πρώτερες εργασίες του πρώτερου έτους για να δει που μπορούν να έγκυται τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουν τη δική τους δουλειά εσωτερικό έλεγχο, ώστε να καταλήξουν σε σωστές επιφυλάξεις. Αυτές οι αιτήσεις, από όταν υπήρχαν αυτές οι αιτήσιες εκθέσεις δραστηριότητα, έχουν εξελιχθεί πολύ και ανταποκρίνονται τι κατευθείαν γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη σύνταξή του. Και όπω τα παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ε, λοιπόν, παίρνουν πολύ καλή, συμμορφώνται πολύ καλά με τι απαιτήσει και για τη διατύπωσή του. Μετά, η μη συνεπή εφαρμογή όμω τη μεθοδολογία για τι ποσοτικοποιημένε επιφυλάξει είναι κάτι παραμένει και το ελεκτικό συνέδριο θα αρχίσει ε, να μην ασχοληθεί περισσότερο με το παλιό, αλλά στο μέλλον να συγκεντρώσει περισσότερε λεπτομέρειες από ό,τι κατά το παρελθόν. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάτι άλλο που αναφέρθηκε σήμερα. Σαν αφορά τι διορθώσει και τι ανακτήσει, εξακολουθούν να είναι τμήμα του προγράμματο ελέγχου όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών. Και εξακολουθούμε λοιπόν να εξετάζουμε το θέμα σύμφωνα με τη συνέχεια που δίδεται. Όσον αφορά τι διακοπέ και αναστολέ, παρατηρούμε ότι σχεδόν το 1-5 φαίνεται να αφορούν τις διακοπές οδήποτε είδους. Όταν ξαναρχίζουν οι πληρωμές, αυξάνεται ο όγκος για το δεύτερο ήμιση των δημοσιονομικών προοπτικών, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει τα προγράμματα. Διότι όλοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τα χρήματα που είχαν διατεθεί στην αρχή. Αυξάνεται λοιπόν ο κίνδυνος σφαλμάτων ετί αυτή η περίπτωση. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά πρέπει να αναστείλεις και να διακόψεις, από την άλλη βλέπουμε ότι ελοχεύουν άλλοι κίνδυνοι που τους γνωρίζει πιστεύω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα μέσα αυτή τη χρηματοπιστωτική μηχανική, Financial Engineering, έκανε κάποια βήματα επιτροπή για να βελτιώσει την υποβολή αναφορών και την ενημέρωση, αλλά γιατί θέλει να επεκτείνει τη χρήση αυτών πριν εφαρμοστούν οι προτινόμενες αλλαγέ Κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Επί σειρά ετών το ίδιο πρόβλημα. Και εδώ ίσως δημιουργούμε ένα τεράστιο νέο πρόβλημα, διότι από οικονομική έποψη ε, ε, ε, η πίστοση, η επαναλαμβανόμενη είναι καλύτερη από μια άπαξ χορηγία. Αλλά δεν γίνεται σωστή διαχείριση, δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι και αν διαδίδονται και πολλαπλασιάζονται. Τέλος, κάτι που δεν αναφέρθηκε σήμερα αλλά στις γραπτές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο είχε αναφερθεί. Συνοχή, ενέργεια και μεταφορές. Σε συγκεκριμένη ε, ε συγκεκριμένο έλεγχο. Δεν είναι τέτοιο ερώτημα, θέλω να το θέσω. Το λεκτικό συνέδριο έχει συνήθεια να αναπροσαρμόζει την ομαδοποίηση ανάλογα με την ανέση κινδύνου που κάνουμε και τα αιτήματά σα. Αυτό είναι απαραίτητο για να παρακολουθούμε τι εξελίξει τη αλλαγή όσον αφορά του κινδύνου του προπολογισμού. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πού βρίσκονται οι κίνδυνοι και να μπορούμε να σας δείξουμε ξεκάθαρα στα πορίσματα του ελέγχου πού είναι αυτοί οι κίνδυνοι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Συνοχή, ενέργεια και μεταφορές έχουν παρόμοια σχήματα ασφαλμάτων. Λοιπόν, σχετίζονται σε μεγάλες υποδομές. Και ο φορέας δεν θέλει να συγχέσει τα δείγματα. Προσπαθούμε να τα εξετάσουμε με έναν συνολικό τρόπο γιατί είναι παρόμοια τα είδη των σφαλμάτων. Αν βγάλουμε ενέργεια και μεταφορές από τη συνοχή, δεν θα αλλάξει το ποσοστό σφαλμάτων από τον τομέα της συνοχής. Ελπίζω αυτό να απαντά το ερώτημα και ελπίζω να μας υποστηρίσει και στο μέλλον η ε, Επιτροπή αυτή, τόσο ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε την ομοδοποίηση των διαφόρων ε, πολιτικών. Σαφές το, Σαφές το μήνυμα, κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. Ακούγονται τόσο πολλές σκέψεις που είναι δύσκολο από πού να ξεκινήσει κανείς εδώ. Αλλά ας ξεκινήσουμε με την προχρηματοδότηση. Δεν ήθελα να επικεντρωθώ σε αυτό στον τομέα της συνοχής. Εγώ είχα σκεφτεί πιο πολύ τον τομέα όπου κάτι μπορείτε να καταφέρετε. Αλλά αν δούμε την προχρηματοδότηση στη συνοχή, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη ε, οδηγεί σε απέτηση για προχρηματοδότηση. Όμως στον τομέα της συνοχής μας δίνει περισσότερο πονοκέφαλο ακόμα, γιατί αυτό για το οποίο μιλάμε είναι ότι πολύ πιθανό τα κράτη-μέλη να μην τηρούν τους κανόνες παρά τους κανόνες. Και μιλάμε για τη διακοπή, την πάυση πληρωμής κτλ. Αλλά είναι εύκολο να λέμε πάυση της προχρηματοδότησης. Τότε κινδυνεύετε να φτάσετε στο κόκκινο. Αλλά από την άλλη μεριά, και εδώ νομίζω ότι έχετε δίκιο, η διακοπή και η πάυση Κοιτάξτε, έχετε διάφορα, έχετε ολόκληρο πλωστάσιο, έτσι. Και αυτό που εμεί θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα, αυτό το πλωστάσιο που διαθέτεται, πώς το χρησιμοποιείτε και πώς αυτό επηρεάζει το ποσοστό σφάλματος. Απ' τη μια έχετε το EDF, όπου σημειώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό διακοπών και από την άλλη μεριά στο κοινωνικό ταμείο έχουμε διακοπή με διαφορετικό ποσοστό σφάλματος. Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο η χρήση των όπλων σας επηρεάζει το ποσοστό σφάλματος στην κάθε περίπτωση. Γιατί στο τέλος η ερώτηση είναι ή έχετε τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα όπλα στη διάθεσή σας αλλά δεν τα χρησιμοποιείτε αρκετά ή δεν έχετε τα κατάλληλα όπλα οπότε πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς θα αποκτήσετε τα όπλα αυτά που χρειάζονται. Γι' αυτό θέλουμε να ξέρουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα δύο μέσα, την ε, διακοπή δηλαδή και την άρση πληρωμών, πώς τα χρησιμοποιείτε. Και στον κύριο Ταβέρν θέλω να ρωτήσω κάτι. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε στην παρουσίασή σας για το πώς αντιμετωπίζετε εσείς τον ε, δημοσιονομικό κίνδυνο και τις εγγύσεις που έχουν να κάνουν με τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Από τη μια λοιπόν ε, με κάνετε να νιώθω καλά ότι όντω ελέγχουμε τα πάντα, πολύ ωραία. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν εσείς είσαστε υπόλογο για τον κίνδυνο τον οποίο γνωρίζετε, όπως λέτε, και δεύτερον ότι δεν πρόκειται για τεράστια ποσά. Από την άλλη όμως, το 67 εκατομμύρια που λέτε. Απ' την άλλη όμως επιβεβαιώνεται ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Και εδώ είναι που θέλω να ξέρω περισσότερο μήπως τελικά αντί να καλυτερέψουν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Επίσης, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει και ένα τεράστιο τραπεζικό λογαριασμό με άπειρα χρήματα. Συνεπώς, ακόμα και μικρά ποσά μπορεί να έχουν μεγάλες επιπτώσεις. Δηλαδή από τη μια μεριά με κάνετε να... από τη μια μεριά με καθησυχάζετε ότι παρακολουθείτε την κατάσταση, υπό έλεγχο, εντάξει, οπότε έχω εμπιστοσύνη σε εσά. Από την άλλη μεριά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ορθά ανοιχτά, γιατί αντί να πάνε καλύτερα τα πράγματα μπορούν να πάνε χειρότερα. Και αν είχαμε άπειρα ποσά στη διάθεσή μας, ένα μεγάλο τροπεζικό λογαριασμό, δεν θα ανησυχούσα, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτές είναι οι σκέψεις μου επί του παρόντος. Και να διευκρινιστεί το θέμα των επιφυλάξεων, ίσως να επανέλθω σε αυτό αργότερα. Δεν ξέρω αν ε, ήταν ερωτήσεις ή ήταν συμπεράσματα αυτά. Ας κρίνουν άλλοι. Ωραία, ας πούμε ότι είναι συμπεράσματα, γιατί η συζήτηση έτσι κι αλλιώς ε, συνεχίζεται και με τους επιτρόπους, ο κύριος Σεμέτα ξανάρχεται και τον κύριο Μποσίκης θα έχουμε με μια έκθεση σύντομα. Οπότε νομίζω ότι η συζήτηση που είχαμε ήταν αρκετά πλήρης με ένα σώρο ερωτήσεις, σίγουρα θα προκύψουν κι άλλες. Οπότε κάναμε ένα παραπάνω βήμα προς την κατεύθυνση της απαλλαγής. Εντάξει, ωραία, κλείνει αυτό το θέμα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας εδώ. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Μπαλτσίτη, για την... και θα έχουμε και παρουσίαση και του Επιτρόπου για την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων. Θα ακούσαμε πρώτα τον Επίτροπο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. So I will try to be... Uh, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος παρουσιάζοντας το θέμα. Χαίρομαι που παρουσιάζω επί τη ευκαιρία την ετήσια έξι Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατά πολέμηση των απατών δυνάμει του άρθρου 325. Έκθεση του άρθρου 325 περιγράφει τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη το 2010 για την πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση ατασταλιών και απατών δίνει στατιστική επισκόπηση όλων των ατασταλιών που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη το 2010, συμπεριλαμβανομένων υποθέσεων όπου υπάρχουν υπόνοιες απάτης. Επίση, παρέχονται λεπτομέρειε για την ανάκτηση των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τελικά, η έκθεση κάνει συστάσει περί τη προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Μπορεί να βελτιωθεί αυτή. Αυτή η έκθεση αφορά ειδικό τμήμα για τον κίνδυνο διπλής χρηματοδότηση στον τομέα των πολιτικών συνοχής. Αυτό αντιστοιχεί στην πρώτερη αίτηση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λεπτομερέστερα στοιχεία στο έγγραφο εργασίας για εφαρμογή του άρθρου 325 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς εφαρμόζεται το άρθρο αυτό από τα κράτη-μέλη. Το έγγραφο αυτό συνοδεύει την έκθεση του χρόνου. Στο τμήμα αυτό θα αναφέρουμε τις στρατηγικές ελέγχου και τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον τομέα τη πολιτικής συνοχής. Θα είναι ένα πρώτο βήμα αυτό για να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για λεπτομερή ανάλυση στρατηγικών και μέτρων που εφαρμόζονται από κάθε κράτος μέλος. Πέρα από το έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σταλίες που κοινοποιήθηκαν το 2010, Υπάρχουν άλλα δύο έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση. Το ένα έγγραφο δίνει λεπτομέρειες συνεισφορά των κρατών μελών στην έκθεση και το άλλο έγγραφο δίνει μια επισκόπηση της συνέχεια που έδωσαν τα κράτη-μέλη στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην προηγούμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τα πορίσματα και τις βασικές στατιστικές τάσεις της εκθέσεως της φετινής, να τονίσω τα εξή. Πρώτον, τα γενικά στοιχεία για το 2010 δείχνουν ότι ο αριθμός των τασταλιών που αναφέρθηκαν έχει αυξηθεί σχεδόν για όλους τους τομείς. Η αύξηση ήταν η μεγαλύτερη στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Εκεί ο αριθμός των υποθέσεων ατασταλιών που αναφέρθηκαν αυξήθηκε στις 7.062 το 2010 σε συγκρίση με 4.737 το 2009. Εκτιμόμενη οικονομική συνέπεια των ατασταλιών αυξήθηκε στα 3,15% όλων των χρημάτων ετέθηκαν στον τομέα το 2010 σε συγκρίση με 2,44% το 2009 η αύξηση στους τομείς της γεωργίας και των άμεσων δαπανών ήταν πολύ μικρότερη. Στους τομείς των πενταξιακών ταμείων και τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους, ο αριθμός των ατασταλιών που αναφέρθηκαν μειώθηκε. Επίσης, η γενική οικονομική συνέπεια των ατασταλιών που εντοπίστηκαν από τα ελεκτικά συστήματα αυξήθηκαν και στον τομέα των δαπανών και στα έσοδα. Βασικοί λόγοι για αυτή την εξέλιξη είναι δύο. Πρώτον, κυκλικός χαρακτήρας του προγραμματισμού των ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, κυρίως το κλείσιμο της, της ε, εφαρμοστικής περίοδου 2000-2006 και δεύτερον γενική ανάπτυξη στον όγκο και ταχύτητα ενημέρωσε τα κράτη-μέλη μετά από την εφαρμογή βελτιωμένου συστήματος ε, διαχείρισης ατασταλιών όπως αποκαλείται. Αυτή η αύξηση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητα ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη. Δεύτερον, να τονίσουμε ότι εκτιμόμενη οικονομική συνέπεια όσον αφορά τις υπόνοιες ατασταλιών από 180 εκατομμύρια που είχαμε το 2009 πήγε στα 478 εκατομμύρια το 2010. Παρά αυτό το γεγονός αυτή τη γενική αύξηση παρατηρούμε ότι τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να αναφέρουν πολύ χαμηλά ποσοστά υπονιών απατών. Προσεκλήθησαν αυτά τα κράτη-μέλη να αναφέρουν τι γίνεται με τα συστήματα ελέγχου τους σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απατών και ατασταλιών. Το τρίτο που πρέπει να αναφέρω αφορά τις ανακτήσεις που έγιναν όσον αφορά το έτος που καλύπτεται. Επετεύχθη πρόοδος. Συνολικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ αχρεωστήτως καταφληθέντων ποσών ανεκτήθησαν το 2010. Όμως, περισσότερες προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν κυρίως στην ανάκτηση των προενταξιακών πόρων. Για τους προαναφερθέντες λόγους δεν μας απασχολεί η γενική τάση της ε, που αναφέρεται στη φετινή έκθεση, όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να επιφέρουμε περαιτέρω βελτιώσεις. Γι' αυτό λάβαμε συμπληρωματικά μέτρα για να βελτιώσουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα ήθελα να αναφέρω τα βασικά μέτρα που πήραμε. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συστήσει όλα τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείριση ατασταλιών, ούτω ώστε να βελτιώσουν περαιτέρω την ενημέρωση και την... Ε, για αυτά τα φαινόμενα. Δεύτερον, υθετήσαμε διάφορε πρωτοβουλίε πολιτική, ε, ενισχύοντα έτσι την καταπολέμηση των απατών. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιημένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση των βασικών κανόνων που διέπουν όλε τι δραστηριότητε Όλαφ που υιοθετήθηκε το 2011 τον Μάρτιο έχουμε μια ανακοίνωση για στρατηγική κατά των απατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μια ανακοίνωση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσω ποινικού δικαίου, ποινικού δικαίου και από διάφορες έρευνες. Προσβλέπουμε στην συνέχιση των καλής και καρποφόρας ε, συνεργασίας με την Επιτροπή ε, Ελέγχου Προπολογισμού και θέλουμε όπως κατά το παρελθόν να συνεργαστούμε και στο μέλλον μαζί σας προς όφελος ε, και συμφέρον των φορολογουμένων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε για την αιτήση αυτή έκθεση σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μπαλτσίτη. Δεν ξέρω αν ζητά κανεί άλλο το λόγο για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μπαλτσίτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ τον Επίτροπο που μας παρουσίασε τις πληροφορίες που αφορούν την ε, καταπολέμηση των απατών. Όταν ασχοληθήκαμε με το προηγούμενο θέμα, υπήρχαν κάποια ζητήματα τα οποία συνδεόταν σε κάποιο βαθμό με αυτή την έκθεση και με το περιεχόμενο της εν λόγω εκθέσεως δεν θα ήθελα να χρονοτριβήσω αναφερόμενος στα στοιχεία που ανέφερε ο Επίτροπος και επί των λεπτομεριών. Ε, θα ήθελα να εκφράσω ποια είναι η δική μου πρακτική εμπειρία επί του θέματος. Εάν βασιστούμε σε βραχυπρόθεσμη προπτική, εν τη αυτή περιπτώση, όπως έλεγε και ο Επίτροπος, διαπιστώνουμε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως, το 2012 πιστεύω ότι θα επανέλθουμε στα ίδια θέματα και στα ίδια προβλήματα. Πρώτα απ' όλα διότι τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν δώσει αξιόπιστες πληροφορίες. Από την άλλη πλευρά οι πληρωμές που τα χρήματα που θα προέρχονται από ανακτήσεις δεν θα φτάνουν το αναμενόμενο και το φιλόμενο ύψος. Από την άλλη πάλι τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν εφαρμόσει τους νόμους καταλήλως και ίσως 2 δισεκατομμύρια ευρώ τελικά να μην ανακτηθούν το 2012. Γιατί το σύστημα είναι έτσι που είναι. Διότι όταν τα νέα κράτη-μέλη ε, ήταν στη διαδικασία ένταξης προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχαν πολύ αυστηρές απαιτήσεις για τη χορήγηση κοινοτικών ενισχύσεων και οι χώρες αυτές προσπαθούσαν να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια το έκαναν βασιζόμενα επί στατηγικών προσανατολισμών που ίσχυαν τότε και επί του οράματος που είχαν τα ίδια τα κράτη. Τα κράτη. Και δεν υπήρχε ομοιογένεια. Και δεν υπάρχει ομοιογένεια στον τομέα. Και στις διάφορες χώρες υπάρχουν διαφορετικά συστήματα και χρειάζεται μια βούληση προς μια ομογενοποίηση. Θα καταλαβαίνει ο Επίτροπος πολύ καλά ότι δεν είναι πολύ καλή η κατάσταση και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η κατάσταση και μάλιστα να αλλάξει σύντομα. Σήμερα, τώρα, είναι και η ώρα να δράσουμε, να κινηθούμε. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί δεν ανακτούμε ποσά τόσο μεγάλα. Όταν πέρσι προσπαθήσαμε να δούμε γιατί το ποσοστό απορρόφησης είναι τόσο χαμηλό, είδαμε ότι δεν είχαμε τι αναγκαίε πληροφορίε για να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα. Σήμερα έχουμε τις πληροφορίες της απαιτούμενες. Όσον αφορά την έκθεσή μου, που θα παρουσιάσω σύντομα, εκεί, σε αυτή θα αναφέρω κάποια πράγματα, κάποιες διατάξεις, κάποιους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ανάληψη των ευθυνών. Τώρα τα κράτη-μέλη ουσιαστικά είναι τα μόνα υπεύθυνα για τις ατασταλίες και για τα ποσά που θα έπρεπε να καταβληθούν, που θα έπρεπε να ανακτηθούν και δεν ανακτήθηκαν. Θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι υπεύθυνη για αυτό το θέμα. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη, εν τη αυτή περιπτώσει, θα μπορεί να απαιτεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη χορήγηση πληροφοριών από πλευράς κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι πρέπει να παρουσιάζουν περισσότερες πληροφορίες και από τη στιγμή θα γίνει αυτό να δίνουν περισσότερες πληροφορίες τα κράτη-μέλη τα στατιστικά τους στοιχεία ε, δεν ξέρω αν θα είναι τα θα υποστούν κάποιες πιέσεις. Αλλά άμα θέλουμε να δούμε πιο ξεκάθαρα την κατάσταση, βλέπουμε ότι όσον αφορά τα στοιχεία υπάρχει πρόβλημα από πλευράς κρατών μελών και στατιστικών υπηρεσιών κρατών μελών. Δεν δίνουν επαρκείς πληροφορίες. Είναι θέμα λοιπόν ευθυνών αυτό. Και ποιο αναλαμβάνει τι ευθύνε. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά θα έχει αυτή την ευθύνη, θα μπορέσουμε ε, να βελτιώσουμε το σύστημα, θα είναι πιο εύκολο το πράγμα και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Επιτροπή Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για όλου ήταν πιο εύκολο αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Απ' την άλλη, εδώ και μερικέ μέρε ε, μίλησα με τον επικεφαλής της Όλαφ. Η Όλαφ διαθέτει υπηρεσίες που συλλέγουν στοιχεία όσον αφορά τις απάτες, τις ατασταλείς. όμως εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Η ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και θα επαναλάβω ίσως αυτά που ήδη είπα, αλλά θα ήθελα να πω ότι στη Λιθουανία υπάρχουν πέντε διαφορετικές δομές για τη συλλογή των ιδίων πληροφοριών. Το η Διεύθυνση Ασφαλείας, ο φορέας υπεύθυνο για, για οικονομικά εγκλήματα, η εφορία, οι τελωνιακές υπηρεσίες, όλοι αυτοί οι φορείς που είναι διαφορετικοί, έχουν τράπεζες δεδομένων διαφορετικές και δεν συνεργάζονται απαραίτητα μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μοναδική ε, περίπτωση που ισχύει μόνο στην Λιθουανία. Νομίζω και στις άλλες χώρες υπάρχουν παρόμοια πράγματα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες ούτως ώστε η Όλαφ να μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που ε, διαθέτουν οι φορείς που προανέφερα. Αυτό θα επέτρεπε, αν γινόταν, στην Όλαφ να μπορεί να επαληθεύσει τα διαθέσιμα στοιχεία, να έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και εν αυτή περιπτώση η Όλαφ θα μπορούσε να θέτει περισσότερα ερωτήματα προς τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί τα διδύν ε, πληροφορία αποσιωπήθηκε. Ούτω καθεξής. Γιατί δεν καταφέρνουμε να ανακτήσουμε τα οφειλόμενα ποσά. Όλα τα κράτη-μέλη είναι δημοκρατικά κράτη και όλα θα έπρεπε να λειτουργούν καλά. Όμως τα δικαστικά συστήματα διαφέρουν και τα δικαστήρια σε εθνικό επίπεδο δεν κάνουν όλα όσα θα έπρεπε να κάνουν σε αυτές τις υποθέσεις. Όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης και τις θετικές αλλαγές στον τομέα αυτό, αυτές θα μπορούσαν, οι θετικές, θετικές εξελίξεις θα μπορούσαν να επιταχύνουν την όλη διαδικασία όταν αναφερόμαστε στον εξυγχρονισμό του συστήματος δημοσίων αγορών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει ψηφίσει τις βασικές αρχές. Όμως είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου συστήματος το ταχύτερο δυνατόν. Τα κράτη-μέλη ήδη έχουν κάποια εμπειρία όσον αφορά τις δημόσιες ε, προμήθειες και θα πρέπει και σε αυτό το τομέα ο ανθρώπινος παράγοντας να μειώσει την επιρροή του, να μειωθεί αυτή η συνιστόσα και να εφαρμόσουμε και σύστημα πληροφορικής. Αυτό θα βελτίωνε σημαντικά την όλη κατάσταση και θα διευκόλυνε τη ζωή εκείνων που χρησιμοποιούν τα κοινοτικά χρήματα. Θα ήθελα να πω ότι είμαι υπέρ των διατάξεων που αφορούν τον κανόνα του 50% στον τομέα της γεωργίας. Πιστεύω ότι αυτός ο κανόνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους τομείς όπου χρησιμοποιούνται κοινοτικά χρήματα, επί παραδείγματα, παραδείγματι ε, διαθετικές ενισχύσεις στο Ταμείο Συνοχής. Ίσως θα μπορούσαν να βραχυνθούν και οι προθεσμίες ε, δύο και τέσσερα χρόνια αντί για οκτώ θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα έπρεπε επίσης στο μέλλον να καθορίσουμε επακριβώς τις αρμοδιότητες της Όλαφ. Η Όλαφ έχει το δικό της σύστημα, το δικό της σύστημα για να καθορίζει και να εντοπίζει τις ατασταλίες και εμείς από την πλευρά μας ε, οφείλουμε να καθορίσουμε ξεκάθαρα τους κανόνες ανάκτησης των οφειλωμένων ποσών σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και σε κοινοτικό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Μπαλτσίτης. Δύο άτομα στήσωσαν το λόγο, η κυρία Γκρέσλα και ο κύριος Σκυλακάκης. Κανείς άλλος? Η κυρία Γκρέσλα λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω κι εγώ κάποιες ερωτήσεις για πράγματα που δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Καταρχάς, στην ε, έκθεση αναφέρεται ότι έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ατασταλιών και αυτό αποτελεί επιτυχία. Σύμφωνο. γιατί είναι καλό το ότι αναφέρονται. Αλλά αναφέρεται στη συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται γιατί μειώνεται ο αριθμός των ατασταλιών. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνάδει το ένα με το άλλο. Διευκρινίστε μου παρακαλώ για τις ε, προνταξιακές επιδοτήσεις. Χαιρόμαστε με αυτά που ανέφερε ο κύριος Βαλτσίτης σε ό,τι αφορά την Τουρκία, τη Λιδονία, τη Σλοβενία και το καθεξής. Στην ε, συνοχή έχουμε το ποσοστό ε, ανάκτησης περίπου 20% για την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Πώς εξηγούν οι χώρες αυτές αυτή, αυτό το χαμηλό ποσοστό και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αυξήσει το στο αυτό. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές. Όποιος δεν πληρεί τους κανόνες δεν παίρνει τα χρήματα. Καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω μάλλον πολύ απλά γιατί επιμένουν τόσο πολλά προβλήματα στον τομέα αυτό. Για το σύστημα τώρα, για το τι πρέπει να περιλαμβάνεται στι αναφορέ. Υπάρχουν το καθαριστικό σύστημα, ερώτημα του ποιο σύστημα θα ακολουθηθεί. Αναφέρεται από τη συνοχή ότι κατά την δημοσίευση της έκθεσης υπάρχουν ακόμα πόσα εκκρεμή. Ισπανία, Ιρλανδία, Γαλλία. Τι γίνεται λοιπόν με τις χώρες αυτές. Γιατί είχε διατυπωθεί ένσταση και καταγγελία ότι δεν ε, συμμετέχουν όπως θα έπρεπε να συμμετέχουν. Από τις 29, Σεπτεμβρίου, τι γίνεται, υπάρχει κάποια πρόοδος, υπάρχουν μέσα. Τρίτη ερώτηση ήταν αυτή. Τέταρτη ερώτηση για τις χειρουργικές δαπάνες. Γαλλία, Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι χώρες που έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό υποπτών, ε, υποπτών υποθέσεων. Έχει να κάνει αυτό με το πόσο συχνές είναι οι αναφορές. Γιατί θα θέλαμε πιο πολλές λεπτομέρειες στον τομέα των γεωργικών που είναι πιο απλό να διαπιστωθούν οι ατασταλίες για τη βάση δεδομένων τώρα. Ένα δημιούργημα του Κοινοβουλίου από το 2007. Γίνονται διαπραγματεύσεις για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Για την Όλαφ, συγγνώμη. Που εξετάζουν ακριβώς ποιος θα χορηγεί τα στοιχεία στη βάση δεδομένων αυτή. Ως τώρα αυτό γινόταν από τα κράτη-μέλη. Ποιε είναι οι εμπειρίε που έχετε συλλέξει ω τώρα, ε, Ευχαριστώ, κύριε Κυλακάκη. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε βελτίωση και εντοπίζουμε τις ατασταλίες. Κάτι το οποίο οφείλεται είτε σε κυκλική φύση, είτε σε καλύτερη διαχείριση. Συμφωνώ ότι υπάρχει κάποια πρόοδος, όμως η πολιτική μου παρατήρηση είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως δεν είμαστε στην κατάσταση που βρισκόμασταν πριν το 2010 και 2011 εξαιτίας της περίοδου λιτότητας μέσα στην οποία μπαίνουμε. Το επίπεδο ανοχής λοιπόν των πολιτών μας έχει αλλάξει πολύ και έχει αλλάξει τόσο στις ισχυρές οικονομίες που πληρώνουν για να βοηθήσουν τους άλλους, αλλά και στις πιο αδύναμες οικονομίες όπου διαπιστώνουμε ότι ισχύει πολύ σκληρή λιτότητα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Το επίπεδο του τι μπορούμε να κάνουμε έχει επίσης αλλάξει όσον αφορά τις προσπάθειες καταπολέμησης της απάτης. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι βασιζόμαστε κυρία στα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη δεν χειρίζονται ομοιόμορφα την κατάσταση. Δεν χρησιμοποιούν όλοι την ίδια μέθοδο ή δεν κάνουν όλοι τις ίδιες προσπάθειες. Άρα πολλά πράγματα δεν μετρώνται. Λέτε βελτιώσαμε, δεν βελτιώσαμε, ναι, αλλά κατά πόσο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε καλά μέσα για να μετρήσουμε αυτές τις αλλαγές. Οπότε δεν μπορούμε τελικά να πούμε συνολικά αν υπάρχει βελτίωση, επιδίνωση στον τομέα αυτών, κατά πολεμιστής απάτης. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες και περισσότερες πρωτοβουλίες λοιπόν σε αυτόν τον τομέα. Πρωτοβουλίες και προσπάθειες που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, λέω από την Επιτροπή τα χρειαζόμαστε γιατί η κατάχρηση του ευρωπαϊκού χρήματος δεν είναι καθόλου καλό ούτε για τις χώρες οι οποίες κάνουν κακοδιαχείριση, ούτε για τους πολίτες ε, των χωρών αυτών. Και σας το λέω ερχόμενος από μια χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα. Ότι είναι κάτι που άλλαξε τη στάση του κόσμου απέναντι στη δημόσια ζωή. Και το πώς χειριζόμαστε τα δημοσιονομικά ζητήματα. Συνεπώς, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Τώρα, ο Επίτροπος για να απαντήσει παρακαλώ. Πολλές οι ερωτήσεις, ίσως κάποιες να θέλετε να τις απαντήσετε γραπτά, αλλά πάντως ό,τι μπορείτε να μας απαντήσετε τώρα, σας ακούμε. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος, θα προσπαθήσω να απαντήσω, να συνοψίσω. Έρχομαι στις ε, ερωτήσεις που θέτει ο εισηγητής πρώτα απ' όλα. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ποιος έχει την ευθύνη γιατί. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό εδώ να μην ε, μπερδεύουμε τις ευθύνες και να μην λέμε ότι όλες ε, οι ευθύνες περνάνε στην Επιτροπή ενώ τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι. Καταρχήν, είναι ευθύνη των κρατών μελών, μια που πρόκειται για κοινή διαχείριση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι γίνεται ορθά η δαπάνη των κονδυλίων. Αυτά προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση, αυτό είναι ο νόμος και αυτό πρέπει να κάνουν. Και θα είμαι αυστηρός. Το έχω ήδη πει στα κράτη-μέλη που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, το έχω πει. Αλλιώς, δεν γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπλοκη. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά των κρατών μελών. Πρέπει να ξέρουμε από τα κράτη-μέλη τι γίνεται. Το μεγάλο βάρος λοιπόν της ευθύνης πρέπει να είναι στο επίπεδο των χωρών μελών. Βέβαια, βελτιώσεις πάνω στις οποίες δουλεύουμε, ο κανονισμός της Όλαφ για παράδειγμα, όπως τα είπε και η κυρία Γκλέσσελ, η νέα στρατηγική καταπολέμηση της απάτης, όπου ζητάμε από όλες τις γενικές διευθύνσεις να αναπτύξουν τη δικιά του στρατηγική καταπολέμηση της απάτης, είναι θετικά βήματα ή και από πλευράς της πρόληψης της απάτης. Γίνονται λοιπόν πράγματα τα οποία πιστεύω ότι θα αποφέρουν καρπούς. Του χρόνου θα έχουμε και νομοθετική πρόταση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Πρόθεσή μας είναι, ποινικά δηλαδή, πρόθεσή μας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα θα ενισχυθεί, πιστεύω, η ευθύνη των κρατών μελών. Όσον αφορά την νομοθετική δουλειά, προχωράμε σημαντικά και πιστεύω ότι και ελπίζω ότι οι προτάσεις αυτές που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκριθούν από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνεπώς, για τα χαμηλά επίπεδα ίσπραξης. Πρέπει να σας πω, όταν πηγαίνω στις χώρες μέλη, συζητάω και δεν συζητάω μόνο, το λέω και δημόσια, ότι υπάρχουν προβλήματα με την ίσπραξη. Έτσι δημιουργείται κάποια πολιτική πίεση. Στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία για παράδειγμα όταν πήγα, το είπα και δημόσια. Η Όλαφ από την πλευρά της φυσικά και επιμένει και πιέζει για την ίσπραξη. Αλλά υπάρχουν πρακτικά ζητήματα με την ίσπραξη γιατί τα χρήματα δαπανώνται σε επίπεδο δικαιούχων και δεν είναι πάντα τόσο προφανές να πάρει κανείς πίσω τα χρήματα να τα εισπράξει, γιατί μερικές φορές οι δικαιούχοι έχουν πτωχεύσει. Οπότε πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά. Και γι' αυτό μερικές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις. Για αντικειμενικούς λόγους. Αλλά όταν ε, δεν πρόκειται για αντικειμενικούς λόγους, τότε πρέπει, και το κάνουμε, πιέζουμε τις χώρες μέλη. Για το θέμα των συστημάτων διαχείρισης των ατασταλιών και των ε, συστημάτων που υπάρχουν στην έκθεσή μας και που μένει να εφαρμοστούν από τις πληροφορίες που έχω, όλα αυτά τα συστήματα ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Συνδέονται με το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι από του χρόνου θα αρχίσουν να αποφέρουν. Θα χρησιμοποιείται δηλαδή το νέο σύστημα. Φυσικά και πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητα με διάφορα υποπρογράμματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το λέμε. Το πολύ χαμηλό επίπεδο αναφερομένων ατασταλιών και απατών ή υπονιών που υπάρχουν για απάτες έχει σαν αποτέλεσμα να σκεφτόμαστε μήπως κάτι πάει στραβά με το σύστημα και μήπως γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πιο πολύ τις περιπτώσεις των χωρών εκείνων που αναφέρουν ε, πολύ χαμηλό επίπεδο ατασταλιών ή απατών. Για μένα το υψηλό επίπεδο είναι εκείνο του σφάλματος που εντοπίζει τελικά το ελεγκτικό συνέδριο. Όταν συζητούσαμε το προηγούμενο σημείο, είδατε ότι το ελεγκτικό συνέδριο κάνει εκτιμήσεις βασίζει τα στοιχεία του όχι μόνο στις συγκεκριμένες εκθέσεις αλλά και στην εκτίμηση που κάνουν. Οπότε ιδεοδός τα, ποσά, τα ποσοστά, μάλλον τα επίπεδα ατασταλιών πρέπει να είναι πολύ κοντά στο επίπεδο σφάλματος που εντοπίζεται τελικά από το λεκτικό συνέδριο. Γιατί τότε σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη όντως αναφέρουν όλα όσα υπάρχουν και συμβαίνουν στη χώρα τους. Όταν ταυτίζονται τα δύο επίπεδα είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Ποια ήταν η τελευταία ερώτηση. Τη βάση δεδομένων. Η Όλαφ χρησιμοποιεί κυρίως την διαχείριση, το σύστημα διαχείρισης ατασταλιών. Δεδομένα δηλαδή τα οποία τροφοδοτούν ε, την Όλαφ και έρχονται βάσει της περιγραφής η οποία υπάρχει σε αυτό το σύστημα διαχείρισης ατασταλιών. Μόνο στην προένταξη Ε, έχουμε γραπτές εκθέσεις. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Στόχος μας είναι να περάσουμε στην ηλεκτρονική αναφορά και μεταφορά δεδομένων. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής τώρα έχει το λόγο, ο κύριος Μπαλτσίτης, για να κλείσουμε αυτό το σημείο. Mm. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ανοιχτός, απαντώντας όλες τις ερωτήσεις, κυρίως όσον αφορά την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υποβάλω τις προτάσεις μου, θα δω ποια είναι η γνώμη των συναδέλφων, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά της στον τομέα της κατά πολεμήσεως των απατών, τα ίδια δικαιώματα που διαθέτει και στον τομέα του ανταγωνισμού. Ε, για συγκεκριμένη και μια συγκεκριμένη υπηρεσία όπως η Όλαφ θα μπορούσε να λάβει την εντολή να διενεργεί έρευνες, να συλλέγει έγγραφα κλπ βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα πρόθυμα να δίνουν τι αναγκαίε πληροφορίε. δεν δίνουν όλα όσα πρέπει και θα ήθελα να ζητήσω να καθυστερήσει η παρουσίαση της εκθέσεώς μου διότι πρόκειται περί σημαντικότητα του εγγράφου, θα έπρεπε να το υποβάλω κανονικά στις 4 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και είναι δύσκολη περίοδος και αν είναι δυνατόν θα ήθελα να εξετάσουμε την έκθεσή μου αργότερα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες καλές χριστουγεννιάτικες διακοπές και ελπίζω στο μέλλον όλοι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την απάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα. Ευχαριστώ. So, thank you. Yeah, still you have meeting. Uh, thank you. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μπαλτσίτης και θα κοιτάξουμε τι γίνεται με την προθεσμία για την κατάθεση της έκθεσής σας. Θα θέλαμε να τη συζητήσουμε στις 24 Ιανουαρίου επί της αρχής και βιαστήκατε να μας ευχηθείτε καλά Χριστούγεννα γιατί έχουμε άλλη μια συνεδρίαση που ελπίζω να δω πολλούς συναδέλφους όπως και να έχει. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που έμεινε όλο το πρωί μαζί μας για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε, να ευχαριστήσω και τους ε, βοηθούς του, τους ε, συνεργάτες του για όλη τη βοήθεια και θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Να περάσω στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα το πρωί, στο 6, παρουσίασε της έκθεση της ε, επίσκεψής μας με την αντιπροσωπεία στο Κανταράς, όπου έχει την έντρα του το πρόγραμμα ITER στη Γαλλία. Έχετε όλα τα στοιχεία, όλα τα έγγραφα στην διάθεσή σας. Στη σελίδα 11 και 12 στην αγγλική έκδοση βλέπετε τα συμπεράσματα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων και ήταν κοινή επίσκεψη μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού, ε, αξιολόγησαν θετικά, αρκετά θετικά το πρόγραμμα του ΙΤΕΡ και θεωρούν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και ότι η χρηματοδότησή του δεν θα πρέπει να διακοπεί ή να ανασταλεί. Αλλά ότι όλα αυτά θα πρέπει να συμβούν υπό κάποιες πολύ συγκεκριμένες συνθήκες διαφάνειας, επαρκούς ελέγχου των αποφάσεων, ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης, ε, εκ νέου αξιολόγηση του κόστους, υποβολή εκθέσεων σε τακτικά διαστήματα για τις ε, ανάγκες του έργου, διαφάνεια και έλεγχος ε, σε ό,τι αφορά τα έγγραφα εσωτερικού ελέγχου. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν μπορείτε να τα διαβάσετε. Η μεγάλη λοιπόν πλειοψηφία των συναδέλφων αξιολογούν και εκτιμούν θετικά τα όσα είδαμε επί τόπου. Μία επιφύλαξη διατυπώθηκε από τους πράσινους και από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά και από τις πράσινους ε, από τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία ήταν ε, θετική και έχουν ληφθεί και ε, μέτρα από την Επιτροπή Προπολογισμού για την περαιτέρω χρηματοδότηση για το, την περίοδο 2012-2013. Ε, δεν ξέρω, έχετε ερωτήσεις, έχετε διευκρινήσεις που θέλετε να σας δώσω ή θέλετε, θεωρείτε ότι μπορούμε να εγκρίνουμε το σχέδιο αυτό. Όλοι συμφωνείτε. Πολύ ωραία. Άρα αυτή θα αποτελεί και την επίσημη έκθεση σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στο Καταράσου. Η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται για τις 19 και 20 Δεκεμβρίου. Ζητώ ρητά να επιδείξετε κάποια πειθαρχία και να παραστείτε. Γιατί έχουμε σημαντικά θέματα να συζητήσουμε και με σημαντικούς ε, προσκεκλημένους. Την τελευταία φορά που ο κύριος Μάιστατ... Είναι η τελευταία φορά που θα έρθει ο κύριος Μάιστατ από την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί συνταξιοδοτήθε και θα αντικατασταθεί. Άρα σας παρακαλώ στις 19 και 20 του μηνός να παρευρεθείτε όσο πιο πολύ πολύ αριθμή γίνεται. Αν δεν έχετε κάτι στα διάφορα να κλείσουμε και να ζητήσω όσους δεν έχουν δουλειά να κάνουν στα πλαίσια της συνεδρίασης των συντονιστών να εξέλθουν τις αιθούσεις το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου και κλεισμένων των θυρών να διεξαχθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ.